Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ Εξωτερικών της Γκάνα, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί κύριοι βουλευτέ. Κυρίε και κύριοι πρεσβευτές, κύριε και κύριοι τα παιδιά, μόλι πριν από 30 χρόνια στι 20 Νοεμβρίου του 1989 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε ομόφωνα τη νέα διεθνή συνθήκη δεσμευτική νομικά που σήμερα παραμένει η διεθνή συνθήκη που έχει επικυρωθεί από τα περισσότερα κράτη-μέλη. αφορά τους ε, ανηλίκους σε σχέση με την αναγνώριση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων μετά από δεκαετίες αγώνα και υπομονής κατάφεραν ε, πολλές άντρες και γυναίκες που δώσαν αυτόν τον αγώνα να αλλάξουν την νοοτροπία, να παρακάψουν τις παραδόσεις για να θεσπίζουν νέους κανόνες για να εγγυηθούν ότι ποτέ οι ανήλικοι δεν θα θεωρηθούν ξανά η διοκρισία των γονέων ή των ενηλίκων ή οποιασδήποτε άλλης ε, αρχής και αυθεντίας αλλά ότι θα είναι ανθρώπινα όντα με τα δικαιώματά τους τα οποία γίνονται σεβαστά και προστατεύονται και το ότι συνεδέθησαν στο πρόσωπο του ανηλίγου αυτό δεν ήταν κάτι αυτονόητο. Οπότε γι' αυτό και θα πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς τους οξυδερικείς άντρες και γυναίκες με τόση γενεοδορία και έλτουριστές. Χωρίς αυτούς δεν θα είχε γίνει ποτέ αυτή εδώ η εκδήλωση. Οι ανήλικοι επλήγησαν από ακραία φτώχεια μετά τον πρώτο ε, Παγκόσμιο Πόλεμο η Έγκλεντα Εντζέμ από την Βρετανία κατήρτισε έναν χάρτη το 1924 εκεί όπου ενσωματώνονται τα βασικά δικαιώματα των Ελλήνων αυτή την οποία τη διαβίβαζε στην κοινότητα των εθνών. Η δε διακήρυξη της Γενέβης ε, από όπου βγήκε αυτή, ε, αυτή η χάρτα έθεσε τα πρώτα νομικά διεθνή θεμέλια δεν ε, ήταν ε, δεσμευτική ε, αυτή η διακήρυξη όλα αυτά παραμένει στο ένα ιστορικό έγγραφο και ο Πολωνός Πέτρος Γιάννους Κόρτζακ στον δεύτερο παγκοσμίο πόλεμο τη χρησιμοποίησε για την προστασία των ανηλίκων και διακήρυξε από την αρχή την προστασία τους από την βία του πολέμου και ε, υπήρχε το δικαίωμα στη ζωή πίστηκε ε, η απόλυτο σεβασμός ε, στην παιδική ηλικία και η Γκεστάπο τον συνέλαβε και άφησε τελευταία του πνοή στο στρατόπεδο συγκέντρωση της Τριμπλίνκα το 1942 κρατώντας τα παιδιά κοντά του και η χώρα του η Πολωνία πρόκειται να υιοθετήσει αυτό τον αγώνα και το 1979 πρότεινε στην Γενική Σύνδεση του ΟΗΕ να καταρτήσει αυτό το δεσμευτικό κίνημα για τα κράτη και αυτό να ενσωματωθεί στην Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 ως, ε, και, και επίσης ε, και στην ε, δήλωση για τα δικαιώματα του παιδιού του 1959. Οπότε χρειαστήκαν 10 χρόνια σκληρής δουλειάς. Και έτσι είχαμε τον κωδικοποίηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχουν σχέση με τους ανηλίκους των, τους κάτω των 18 ετών και αυτό και σήμερα τιμούμε στις 20 Νοεμβρίου ε, την ε, Παγκόσμια Μέρα για τα παιδιά και οπότε τώρα έχουμε αυτόν τον παγκόσμιο πυλώνα ο οποίος στηρίζει τα δικαιώματα τα σημαντικά και απαραίτητα ούτως ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν πλήρως οι ανήλικοι και επίσης έχουμε αυτό το ανθρωπιστικό σύμβολο ε, το οποίο το εκπροσωπούν πάρα πολλές οργανώσεις που πασχίζουν για τα δικαιώματα των ανηλίκων σε όλο τον κόσμο και έχουμε επίσης και ένα νομικό πλαίσιο των οργάνων του ΟΗΕ, UNICEF και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Επίσης, ε, ε, αυτό πρόκειται να είναι μια ε, σημεία πολιτική για τα κράτη, τα οποία έχοντας προσχωρήσει στην συνθήκη έχουν δεσμευτεί να τηρήσουν τις σχετικές υποχρεώσεις και δέχονται να είναι αντικείμενα ελέγχου και δημόσιας αξιολόγησης. Το πρώτο κράτος στον κόσμο το οποίο κύρωσε αυτή τη συνθήκη είναι η δημοκρατία της Γκάνα. Και έτσι ήταν το παράδειγμα προς μίμηση. Σήμερα έχουμε 197 χώρες οι οποίες ακολούθησαν το παράδειγμα της Γκάνα. Μεγαλειώτης Κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, σήμερα συναντηθήκαμε για να ε, τιμήσουμε και να γιορτάσουμε με ενθουσιασμό αυτές τις ε, νίκες που έχουμε πετύχει και έτσι επομένως θα προτάξουμε όλες τις νίκες που ακόμα θα πρέπει να κατακτήσουμε ε, μαζί οι νομοθέτες, οι ειδικοί, τα δημόσια πρόσωπα, ε, όσοι έχουν αφοσιωθεί σε αυτόν τον αγώνα αλλά και οι ανήλικοι. Με τις σημερινές συζητήσεις πρόκειται να βρούμε μια καινούργια διαδρομή. Θα τάξουμε καινούργιες ε, προτεραιότητες ούτως ώστε θα αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις ε, του καιρού μας που έχουν σχέση με την ανάπτυξη το μεγάλωμα του παιδιού την εποχή του, της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιακής ε, τεχνολογίας είναι απαράδεκτο ακόμα να πεθαίνουν ε, κάθε χρόνο περισσότερα από 6 εκατομμύρια ε, ε, ανήλικοι με ηλικία κάτω των 15. Αυτό σημαίνει ότι πεθαίνει ένα παιδί κάθε 5 δευτερόλεπτα. Συνήθω αυτό θα μπορούσε να αποφευθεί. Πάντω, σύμφωνα με τις ε, εκτιμήσεις, εάν ταχαίω να λάβουμε δράση θα έχουμε πάνω από 55 εκατομμύρια ε, από παιδιά κάτω των 5, τα μισά από τα οποία θα είναι νεογέννητα, τα οποία πρόκειται να πεθάνουν μέσα στο 2030. Είναι αδιανόητο ναι, πάνω από 152 εκατομμύρια παιδιών να στερούνται της παιδικής τους ηλικίας και της ε, εκπαίδευσης διότι δουλεύουν σε εργαστήρια, σε ε, εργοστάσια, σε ορυχεία χωρίς να αναφέρουμε το πόσο τα εκμεταλλεύονται. Πρόκειται για δουλεία, ε, εκπόρνευση, για στατολογισή τους στους πολέμους. Τώρα που μιλάμε γίνονται όλα αυτά και τον περασμένο μήνα ο ΙΕ επισήμανε στα κράτη-μέλη ε, το τι ισχύει όσον αφορά αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν στερηθεί τη ελευθερία τους πάνω από 1,5 εκατομμύριο βρίσκονται φυλακισμένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουν επαφή με τον εξωτερικό κόσμο. Πρόκειται για τρομακτικά νούμερα τα οποία μας συγκλονίζουν και που αντιστοιχούν σε όλα αυτά τα χαμόγελα τα οποία έχουν κλαπεί από τα παιδιά στην αθότητα που έχει χαθεί και με την ευκαιρία που η νέα του Κοινοβουλίου μας προσφέρει θα πρέπει να εκπονήσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, θα πρέπει να καθορίσουμε ξεκάθαρους στόχους για την επόμενη πενταετία. Το Κοινοβουλίο επίσης ε, τώρα συντάσσει ένα ψήφισμα το οποίο πρόκειται να εγκριθεί την επόμενη εβδομάδα και αυτό θα αποτελέσει υλικό για, για τις δικές σας συζητήσεις. Επίσης θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την νέα πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, τη δήλωση ότι θα αφοσιωθεί στην προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων και ότι πρόκειται για πολιτική της προτεραιότητα. Και είμαι βέβαιος ότι σε αυτή την προσπάθεια θα την υποστηρίξει πλήρως το Κοινοβούλιο. Και αυτή η διάσκεψη θα πρέπει να θεωρηθεί επίσης μια σημαντική συμβολή στην στρατηγική και τα δικαιώματα των ανηλίκων τα όσα έχουν απασχολήσει την ε, ε, υποψήφια επίτροπο για την ε, δημοκρατία και το δημογραφικό ζήτημα την κυρία Σουίτσα οπότε όλα αυτά θέλουμε να τα προωθήσουμε μέσω της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει κάποια σχέδια, κάποιες προτάσεις που κατατείνουν στην πλήξη αυτών των σκοπών. Επίσης τα τελευταία δύο χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην μεγάλη του πλειοψηφία ε, αφιερώθηκε στην προστασία, στην προώθηση των δικαιωμάτων ε, των ανηλίκων και όρισε μια συντονίστρια για τα δικαιώματα των ανηλίκων. Μία από τους αντιπροέδρους της αντιπρόεδρου του Κοινοβουλίου, την Εύα Κόπατς, ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου. Συμφωνώ με την UNICEF ότι τα δικαιώματα των ανηλίκων είναι στενά συνδεδεμένα με το ζήτημα της υλοποίησης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Άρα θα πρέπει να γίνει ειδική προσπάθεια ούτως ώστε να σταματήσουν οι καταχρήσεις, η εκμετάλλευση των ανηλίκων και να καταπολύνουμε την φτώχεια και να πετύχουμε την βελτίωση για την παιδεία, την προσβασιμότητα επίσης ε, στην σωστή διατροφή και Στι Υπηρεσίε υγεία ευχαριστώ όλου όσου συμμετέχουν στο πάνελ επειδή δέχτηκαν να έρθουν και να μας ε, δώσουν την εμπειρία τους ε, όλους αυτού τον αγώνα και το όραμά τους για ένα δίκαιο μέλλον το οποίο αξίζουν τα παιδιά. Ε, Επίση είναι σημαντικό να ακουστεί εδώ η φωνή όλων αυτών των κυρίως ενδιαφερομένων και ιδίως να ευχαριστήσουμε τον Μπέρεκε, τη Σιόντα, την Μαρία, την Ράνια, τον Ακράτ και θα ήθελα να ενθαρρύνω όλα τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εδώ να λάβουν το λόγο σήμερα εδώ στο ημικύκλιο και κάθε φορά επίσης όποτε τους δίνεται ευκαιρία προς το πρόκειται για το δικαίωμα ε, λόγου, πρόκειται για το δικαίωμα στην συμμετοχή το οποίο έχει ενταχθεί στην ε, ε διεθνή σύμβαση το δικαιώματα του παιδιού ακριβώς όπως ε, πάρα πολλοί από εσά έκαναν για το, την αλλαγή του κλίματος και όλοι εμείς οι νύλοι βουλευρά μας έχουμε νομική και ηθική υποχρέωση αλλά και πολιτική να σας ακούσουμε και επίσης θα πρέπει να σας πω ότι ευχαριστούμε την ε, Μεγαλειοτάτη την ευχαριστούμε για αυτές τις, τις προσπάθειε που εδώ και τόσα χρόνια ε, καταβάλει όσον αφορά την υπόθεση των παιδιών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Έχουμε καλή επιτυχία στι εργασίε μα. Έχετε το λόγο με Excellence. Εξοχότητες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί νέοι, εδώ και αρκετά χρόνια μεταβαίνω επί τόπου ως επίτιμη πρόεδρος, πρόεδρος της UNICEF Βελγίου προασπίστρια το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατά τις επισκέψεις αυτές ανέκαθεν φρόντιζα να συναντήσω τα πιο ευάλωτα παιδιά. Αυτά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους. Αυτά που έχουν υποστεί τα τραύματα του πολέμου. Αυτά που διαβιούν σε απόλυτη εξαθλίωση ή τα παιδιά που πάσχουν από αρρώστιες ή αναπηρίες. Τα παιδιά και οι νέοι σήμερα είναι σε καλύτερη θέση για να κάνουν ακουστές τις ανησυχίες τους και τα προβλήματά τους αλλά ταυτόχρονα είναι και σε καλύτερη θέση να προτείνουν λύσεις για αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να χαιρετήσω όλους ιδιαιτέρως τα παιδιά και τους νέους που αποφάσισαν να λάβουν μέρος σε αυτή τη διάσκεψη και να συμμετέχουν στις συζητήσεις που τους αφορούν άμεσα. Τα ευάλωτα παιδιά που συνάντησα έχουν όπως και εσείς κάποια σχέδια για το μέλλον. Οι φωνές τους και οι προσδοκίες τους λοιπόν θα πρέπει επίσης να ακουστούν. Η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού κατά την υιοθέτησή της πριν από 30 χρόνια αποτέλεσε το αντικείμενο μιας εξαιρετικά ευρείας συνένεσης. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών την κύρωσαν. Η βελτίωση της κατάστασης των παιδιών στον κόσμο είναι σαφώς ένα κοινό μας μέλημα. Η σύμβαση διακηρύσει ότι τα παιδιά έχουν δικαιώματα, όπως όλοι οι άνθρωποι. Αλλά έχουν και κάποια ιδιαίτερα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην υγεία και στην παιδεία. Και έχουν αυτά τα ειδικά δικαιώματα ακριβώς επειδή είναι παιδιά. Δεδομένου του ευάλωτου χαρακτήρα τους, θα πρέπει να τύχουν προστασίας απέναντι στη φτώχεια ή στις συγκρούσεις και απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, εκμετάλλευσης ή βίας. Η σύμβαση αναγνωρίζει επίσης την ελευθερία έκφρασής τους και την ελευθερία της γνώμης τους. Η φωνή των παιδιών λοιπόν μπορεί πλέον να γίνει ακουστή. Αξιοσημείωτη πρόοδος έχει συντελεστεί τα τελευταία 30 χρόνια κατά την θέση σε εφαρμογή της διεθνούς αυτής σύμβασης. Η παιδική θνησιμότητα μειώθηκε κατά το ίμιση. Η πρόσβαση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει γίνει πραγματικότητα για τη μεγάλη πλειοψηφία των αγοριών και των κοριτσιών, ακόμη και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η συχνότητα γάμων παιδιών ε, μειώνεται σταθερά και η παιδική εργασία το ίδιο αλλά 12 εκατομμύρια κορίτσια ακόμη παντρεύονται κατά την παιδική τους ηλικία κάθε χρόνο και δεκάδες εκατομμύρια παιδιών απασχολούνται ακόμη στη γεωργία, στα χωράφια, στα εργαστήρια ή ως οικιακές βοηθοί. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε ακόμη τεράστιες προσπάθειες για να υλοποιήσουμε τους στόχους ε, που θέσπισε η διεθνής κοινότητα το 1989. Αφενός, οι δεσμεύσεις δεν έδωσαν τη θέση τους πάντα σε συγκεκριμένες δράσεις. Αφετέρου, ανέκυψαν και νέες προκλήσεις. Για παράδειγμα, οι επιζήμιες για την υγεία συνέπειες της κλιματικής αλλαγής ή η έξαρση των συγκρούσεων που επηρεάζουν με δυσανάλογο τρόπο τα παιδιά. Ή επίσης τα στρεβλά φορές αποτελέσματα και συνέπειες του ψηφιακού κόσμου, όπως είναι η παρενόχληση στο διαδίκτυο, η, η διείσδυση στην προσωπική ζωή των νέων. Ανέκαθα πέδωσα μεγάλη σημασία στην πρόθεση μιας παιδείας με ποιότητα και για τα κορίτσια και για τα αγόρια. Και επίσης στην υγεία και ιδιαίτερα στην ψυχική υγεία. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, η επόμενη πρόκληση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι αυτή της ποιοτική εκπαίδευσης. Σήμερα, πολλοί άριθμοι μαθητές δεν φτάνουν σε επίπεδο γνώσεων και επάρκειας που να αντιστοιχεί στον αριθμό των χρόνων που πέρασαν στα θρανία. Δεν έχουν προετοιμαστεί για να συνεχίσουν τις σπουδέ τους ή για να βρουν μια θέση απασχόλησης. Οπότε δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στο έπακρο το δυναμικό τους ώστε να γίνουν πλήρη μέλη της κοινωνίας και να διαδραματίσουν το ρόλο που τους πρέπει. Σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, υπερβολικά μεγάλος αριθμός κοριτσιών εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είτε γιατί οι οικογένειές τους δεν το κρίνουν σκόπιμο ή θεωρούν ότι τους χρειάζονται στο σπίτι, γιατί πολύ συχνά τα κορίτσια αυτά τα παντρεύουν σε πολύ μικρή ηλικία. Η ψυχική υγεία είναι μια ουσιώδης συνιστόσα της ε, υγείας και το ίδιο ισχύει και για την υγεία των παιδιών και των εφήβων. Αλλά τα ψυχολογικά προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι νέοι και τα παιδιά πολύ συχνά αγνοούνται, ε, αποκρύπτονται ή παραμελούνται. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για όλα αυτά, ακόμη και οι νέοι μεταξύ τους. Όσοι χρειάζονται βοήθεια θα πρέπει να μπορούν να βρίσκουν ένα ευήκον ους και συμβουλές και φροντίδες κατάλληλες για την, ηλικία τους. Εξοχότητες. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί νέοι, η υιοθέτηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού δεν έγινε μόνο μεγάλες προσδοκίες, αλλά επέφερε και σημαντικές αλλαγές. Από τότε μια γενιά παιδιών έχουν ενηλικιωθεί. Αλλά μόνο μερικά από αυτά κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τις ελπίδες τους και να δουν κάποιες αλλαγές να υλοποιούνται. Για να προχωρήσουμε λοιπόν θα πρέπει να ανακτήσουμε αυτό το πάνδημο ενθουσιασμό που επέφερε τότε στις απαρχές της η Σύμβαση. Τις ε, υποσχέσεις που δώσαμε πριν από 30 χρόνια δεν θα πρέπει μόνο να τις επιβεβαιώσουμε, αλλά κυρίως να τις στηρίσουμε. Σας ευχαριστώ. Μεγαλειοτάτη, Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, θέλω να χαιρετήσω ιδιαίτερα θερμά ε, τους νέους που βρίσκονται εδώ ενώπιόν μας σήμερα. Είναι πραγματική τιμή ευκαιρία που έχω να συμμετέχω σήμερα στην Παγκόσμια ημέρα του παιδιού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου γιορτάζουμε ε, το παρόν και το μέλλον του πλανήτη μας. 30 χρόνια πριν συναντήθηκαν ηγέτες για να δεσμευθούν σε μια ιστορική συμφωνία και δημιούργησαν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σήμερα ακόμα βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά να υποφέρουν ε, φτώχεια, ανισότητα, βία, διακρίσεις. Εκατομμύρια παιδιών κάθε μέρα στερούνται των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων. Το δικαίωμα στο να, να ζουν με τις οικογένειές τους, να πηγαίνουν στο σχολείο, να ε, τους αγαπούν, να είναι ευτυχισμένα, να παίζουν και να έχουν μια ταυτότητα, μια παιδική ηλικία στο κάτω-κάτω. Γι' αυτό σήμερα συγκεντρωθήκαμε όλοι εδώ, κυρίες και κύριοι, και σας ζητώ όλους από εσά που παίρνετε τις αποφάσεις στην Ευρώπη να κοιτάξετε γύρω σας και να αναγνωρίσετε ότι δεν επιτρέπεται να διονύζεται αυτή η κατάσταση. Όπως ε, θα είδατε στο βίντεο κλιπ που έχω γυρίσει πριν από τρία χρόνια με τη UNICEF, η κατάσταση αυτή πονάει υπερβολικά. Θέλω να εγγυηθείτε ότι στις πολιτικές σας αποφάσεις θα έχετε πάντα στο κέντρο τα παιδιά και να αποδεικνύετε καθημερινά ότι εργάζεστε για τα παιδιά, να τα λαμβάνετε υπόψη, να λογαριάζετε στα παιδιά και να προωθείτε τα δικαιώματά τους στη συμμετοχή. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη σε εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.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 Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Για κάποιε εικόνε πρόκειται για ε, κάποια λόγια πολύ σημαντικά για μα, για εσά, αλλά κυρίω για τη διαδρομή που θέλουμε μαζί να κάνουμε. σα ευχαριστώ για όσα κάνετε.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

Welcome. Καλώς ορίσατε, λέει η πρόεδρος. Στα αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά, αγαπητοί, προσκεκλημένοι. Καθίστε. Queridos y Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι μεγάλη μου τιμή να κλείσω την έναρξη αυτού του τόσο ώστε να γιορτάσουμε όλοι μαζί την επέτειο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Μια είναι συνθήκη νεαρής ηλικία, αλλά πάρα πολύ σημαντική. Μόλις 30 ετών. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, με την συμμετοχή της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Επιτροπή Γιούρι, συνεκάλεσαν αυτή την διάσκεψη. Και έχουμε το πρώτο πάνελ το οποίο θα εστιαστεί στην κατάσταση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών. Οι συνάδελφοι τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μετά θα συνεχίσουν ε, την συζήτηση μαζί σας και το θέμα θα είναι όλα όσα γίνονται σε όλο τον κόσμο. Ε, θα μιλήσουμε μόνο για τα παιδιά της ε, Ευρώπης και ε, η κατευθυντήρια γραμμή για αυτό το πάνελ είναι το να συζητήσουμε το τι εγγυήσει θα δημιουργηθούν για όλα τα παιδιά εδώ στις χώρες μας είτε είναι καταγωγής ευρωπαϊκής είτε όχι για όλα τα δικαιώματα που τους απονέμει η σχετική σύμβαση το πώς θα τηρούνται και πώς θα καταγγέλλεται η παραβίασή τους άσχετα από ηθαγένεια ή από τόπο κατοικίας. Πρόσφυγες, απάτριδες, μετανάστες. Όποιος βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαπέται από την κοινωνικη νομοθεσία και όλοι οι ανήλικοι έχουν τα δικαιώματά τους προστατευμένα και βέβαια χρειάζονται τον έχουν πρόσβαση σε αυτή την προστασία γιατί πρώτα πρώτα θα πρέπει τα παιδιά να τα μεταχειριζόμαστε ως παιδιά. Αυτή επομένω είναι η κρυθυντήρια γραμμή, το πνεύμα της Επιτροπής ε, ΛΥΜΠΕ, ιδίως όσον αυτό το έργο μας για το κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Πολιτικής Ασύλου και Μετανάστευσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακάματα προσπαθεί να πιέζει να μιλά για την προστασία των ασυνοδεύτων ανηλίκων μεταναστών. Να υπάρξει ορισμός συστηματικά κάποιου επιμελητή τους και να απαγορεύεται η κράτησή τους. Έχουμε προσπαθήσει επίσης και στο μέτωπο της προστασίας των ανηλίκων όσον αφορά τις ε, νομικές δικαστικές διαδικασίες ιδίως με την οδηγία του 2016 σε σχέση με κάποιου είδους δικονομικές εγγύησεις για τα παιδιά τα οποία είναι υποκατηγορία ή θεωρούνται υπόπτα, φέρονται να έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα ε, στα πλαίσια της ποινικής δικονομίας και προσπαθήσαμε να σταθμίσουμε το τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τα τελευταία 30 χρόνια έναν απολογισμό για να υπάρξει εγγύηση του ότι αυτή η σύμβαση θα ενσωματωθεί θα ενσωματωθεί πλήρω στο κοινωτικό δίκαιο, στι ε, συνθήκε, στην νομοθεσία, στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και στην ομολογία των δικαστηρίων. Ούτω ώστε το περιεχόμενο, που είναι το πιο σημαντικό, να έχει πραγματική επιρροή στην ζωή όλο ένα και περισσότερων ε, παιδιών. Και ποτέ δεν θεωρούμε ότι τα πράγματα είναι τέλεια, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι να προσπαθήσουμε παραπάνω. Η Επίτροπος ε, Γιούροβα πρόκειται να έχει το πιδάλιο σε αυτή την προσπάθεια και θα μας πει ε, τι θα γίνει στο μέλλον και με βάση τις ανακοινώσεις της καινούργιας Πρόεδρου της Κομισιόν για μια καινούργια στρατηγική για την προστασία των παιδιών. Και στη συνέχεια πρέπει να δούμε τι και να υπάρχουν, τι ακόμα απομένει να γίνει, ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε τις διακρίσεις, του φραγμού σε αυτή την απόλαυση των δικαιωμάτων από πλευρά των παιδιών. Ο κύριο Σοφλάχερτη, ο διευθυντής της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα θα αναφερθεί σε αυτές τι προσπάθειε συγκεκριμένα από πλευρά τη υπηρεσία του και στη συνέχεια θα ακούσουμε πλευρά τη κοινωνία των πολιτών. Ε, φωνή θα ακουστεί από την ε, κυρία Κολεροπρέκα, η οποία είναι πρόεδρο τη Eurochild, που θα μα πει για τη συμμετοχή των παιδιών στην κοινωνία και για την απόφαση που πρόκειται να διαμορφώσει το μέλλον του. Παρ' όλα αυτά, σας τονίζω το εξή. Πολύ σημαντικό σήμερα έχουμε συμμετοχή σημαντικών ε, προσωπικότητων ανήλικους που ε, θα μιλήσουν στη διάσκεψή μας και σε αυτό το πνεύμα τους ε, καλόλους τους ανήλικους που είναι εδώ όλα τα παιδιά να μιλήσουν για τα δικαιώματά τους. Επίσης, ο Ακράτη Ράινα και Σιόντα ή Ακράτη Ράινα και Σιόντα που πρόκειται να μας πούν τις ε, απόψεις τους όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών. Τι θα πει να είναι κανείς ε, παιδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην σημερινή διάσκεψη για να γιορτάσουμε την 30η επέτειο της Διεθνούς Σύμβασης και σας ευχαριστούμε από καρδιάς που αποφασίσατε σήμερα να έρθετε εδώ και να μας μιλήσετε. Πολύ σημαντικό. Είναι για μας μια μεγάλη τιμή. Επίσης, πριν προχωρήσουμε στο πρώτο πάνελ, πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Γιούροβα, θα ήθελα να σας πω κάποιες ε, πρακτικές λεπτομέρειες για το πώς σήμερα όλοι μαζί θα δουλέψουμε. Οι ερωτήσεις είναι σύντομες. Κάθε λεπτό μετράει. Μπορείτε να ζητήσετε το λόγο, αλλά θα πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο. και αν χρειάζεται κάποια βοήθεια θα σας βοηθήσει το προσωπικό του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό το χαρτί, αυτή την κάρτα για να ζητήσετε το λόγο. Αν έχετε κάτι σημαντικό να ζητήσετε ή να μας πείτε, παρακαλώ ζητήστε το λόγο. Και όταν έρθει η ώρα για να μιλήσετε είναι πολύ σημαντικό. Κοιτάξτε, έχετε κάποια κουμπιά μπροστά σας, θα πρέπει να πατήσετε το κόκκινο κουμπί ε, για να μπορούμε να δούμε η κάμερα να δει πού κάθεστε στην αίθουσα. Ανάλογα με πώς συζητήσουν το λόγο θα μοιράσουμε και τον χρόνο. Το πιο πιθανό είναι να έχετε ένα λεπτό. Μπορεί να πείτε πολύ σημαντικά σε ένα λεπτό. Εμείς όταν λαμβάνουμε το λόγο έχουμε μόνο ένα λεπτό και είμαι σίγουρη ότι και εσείς θα τα πάτε υπέροχα. Οπότε συμπληρώνουμε το έντυπο, την κάρτα και κατόπιν προσέχουμε να πατήσετε το κουμπί να ξέρουμε που είστε. Καταλάβατε. Ωραία, καλώς ορίσατε. Αρχίζει το πανελκύριο γύρω Γιώργο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Uh, Ευχαριστώ πολύ, ε, Μαϊτέ, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι αγαπητοί φίλοι. Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στον εορτασμό σήμερα τη 30ης επαιτίου της έγκρισης ε, της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Καλωσορίζω επίσης την ευκαιρία που έχω να συμμετέχω με τις νεαρές ε, εδώ φίλες στην Αχράτ, τη Ράινα και τη Σιόντα. Αισθάνομαι πολύ νεότερη από ό,τι συνήθω. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την αίσθηση. Ε, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βλέπει τα παιδιά. Αυτό είναι το βασικό. Και μάλιστα ε, από τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι εκείνη που έχει καιρωθεί περισσότερο. Βεβαίως είναι ένα νομικό εργαλείο, αλλά στόχο έχει να δώσει στα παιδιά την ευκαιρία να ζουν παιδικά χρόνια με ευτυχία και υγεία και να έχουν μια δίκαιη ε, ευκαιρία να πετύχουν τον ενήλικο βίο τους. Να σας πω ε, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θελήσαμε να ενισχύσουμε την προστασία των ε, παιδιών. Πολλά ήδη έχουμε πετύχει, αλλά παραμένουν ακόμα πολλά τα παιδιά ε, τα οποία δεν ε, ενημερώνονται, δεν εκπαιδεύονται, παραμένουν στη φτώχεια και στην πείνα. Είναι πραγματικά σπαραξικάρδιο να μαθαίνουμε τις τραγωδίες των παιδιών στη μετανάστευση και θα πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα για να βελτιώσουμε την κατάσταση παγκοσμίω. Πραγματικά εγώ προσπάθησα πολύ να βελτιώσω την κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πολλές προτάσεις με χρήματα από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό για να βελτιώνουμε την κατάσταση των παιδιών ε, με ε, ξενώνες για παιδιά και ε, με ε, επιμέλεια, με προστασία και να μην τους δίνουμε μόνο στέγη και τροφή αλλά και μια προοπτική στην Ευρώπη. Επίσης εργάστηκα πάρα πολύ για να βελτιωθεί η κατάσταση των παιδιών Ρωμά, όπου σε κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε μια δεινή κατάσταση και από την αρχή της ζωής τους ε, είναι καταδικασμένα να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, γιατί δεν έχουν ποιοτική εκπαίδευση. Και εμείς έχουμε νομικά μέσα και οικονομικά για να το αλλάξουμε. Παρόλα αυτά απομένουν πολλά να γίνουν. Επίσης, κάναμε πολλά για να προωθήσουμε μια δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά, όπως ακούσαμε από την κυρία Παγάσα Ορτουντούα. Οπότε έρχονται σε επαφή τα παιδιά με τη δικαιοσύνη ως θύματα ή ε, ως μάρτυρες ή ε, όταν έχουν επιμέλεια ή διαδικασίες ε, μετανάστευσης θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους και η αξιοπρέπειά τους και ότι οι δικαστικές αποφάσεις βασίζονται στο δίκαιο με συμπόνια και με σαφήνεια δεν θα πρέπει η δικαιοσύνη να είναι άλλη μια τραυματική εμπειρία για τα παιδιά. Επίσης αποφασίσαμε να δώσουμε ιδιαίτερη έφαση στα παιδιά όταν είναι θύματα εγκλημάτων. Ιδιαίτερα ε, έχουν το δικαίωμα σε ειδικέ υποστηρικτικές υπηρεσίες που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες πολύ μικρών παιδιών ή παιδιών με αναπηρίες. Και έχουμε βρει κοινού κανόνες για τη στέρηση ελευθερίας, ε, όχι κράτηση, εναλλακτικά και συγκεκριμένες και γρήγορε διαδικασίες της επίλυσης ε, ενέξεων που αφορούν παιδιά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε επαγγελματίες και έχουμε δώσει χρήματα ε, για την εκπαίδευση των ειδικών έτσι ώστε να έχουν τα εφόδια εκείνα ε, που θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τα παιδιά και να τα συνοδεύσουν σε αυτή την πορεία ε, των παιδιών μέσα από τη δικαιοσύνη. Επίσης υποστηρίζουμε τους ξενώνες για τα παιδιά, φιλικά για τα παιδιά σπίτια με προστασία και σήμερα έχουμε τέτοια κέντρα σε 23 κράτη-μέλη που βοηθούν να βεβαιωθούμε ότι είναι καλύτερα προστατευμένα τα παιδιά που είναι μάρτυρες και θύματα εγκλημάτων. Επίσης προάγουμε το διάλογο με το Φόρουμ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τον περασμένο Απρίλιο συζητήσαμε τις καλές πρακτικές και ευνοούμε τη συμμετοχή των παιδιών στην πολιτική και δημοκρατική ζωή στην Ένωση. Και πρόκειται μάλιστα να γίνει και μια σχετική μελέτη. Όπως γνωρίζετε η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει την 1η Δεκεμβρίου. Σε λίγες μέρες για το μέλλον λοιπόν μπορώ να σας διαβεβαίωσω ότι τα δικαιώματα των παιδιών θα παραμένουν πολύ ψηλά στην ε, ατζέντα της μελλοντική Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να σπάσουμε τον επικίνδυνο κύκλο της παιδικής φτώχειας. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για ε, τους ευρωβουλευτές που ζητούν μια εγγύηση έτσι ώστε κάθε παιδί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες. Θα χρησιμοποιήσουμε τη γεωπολιτική μας θέση θέση ως παγκόσμια εμπορική δύναμη για να προωθήσουμε μια πολιτική μητενική ανοχής για την παιδική εργασία. Τέλος, η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την πρόθεση να εγκρίνει μια συνολική στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μέτρα για να προστατεύει ευάλωτα παιδιά, τα δικαιώματα ε, ε, επιγραμμικά, ε, μια δικαιοσύνη χωρίς βία που να την προλαμβάνει στο μέλλον ως Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα θέλω να ασχοληθεί ε, ιδιαίτερα με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην ψηφιακή εποχή ε, οι σχετικοί χάρτες των Ηνωμένων Εθνών και τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολλέ ευκαιρίε από την ψηφιακή επανάσταση, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά, αλλά είναι και πολλά τα προβλήματα και νέε προκλήσει ε, για την εφαρμογή και την επιβολή των δικαιωμάτων. Α θυμηθούμε ότι όταν θεσμίστηκαν αυτοί οι κανόνε ε, το διαδίκτυο και οι νέε τεχνολογίες δεν ήταν καθόλου τμήμα των ζωών των παιδιών. Σήμερα όχι απλώ είναι τμήμα, αλλά κυριαρχούν καθημερινά. Και πάντα λέω ότι το Facebook δεν θα πρέπει να είναι η μητέρα των παιδιών, ούτε το Instagram ο πατέρας τους. Και επιπλέον, στο Instagram και στον επιγραμμικό κόσμο, τα παιδιά όλο και περισσότερο βλέπουν και πείθονται ότι δεν είναι αρκετά έξυπνα, αρκετά όμορφα, ε, ε, αρκετά ικανά. Υφίστανται ένα μόνιμο ε, εκφοβισμό και υποφέρουν από αυτή την παρενόχληση. Θα πρέπει να το δούμε και αυτό και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε για να βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση και να μειωθεί ο κίνδυνος για τα παιδιά μας. Θα ήθελα κλείνοντας να απευθύνω μια έκκληση στους νέους. Να είστε δραστήριοι, να είστε παρόντες και να τα λέτε δυνατά. Στη χώρα μου, στη τσεχική δημοκρατία, που το 1989 ήταν η Τσεχοσλοβακία, γιορτάσαμε τα 30 χρόνια από τη λεγόμενη βελούδινη επανάσταση. Γι' αυτό φόρεσα και το βελούδινο σακάκι μου. Μπορεί να είναι φροηδικό και αυτό. Άρχισε λοιπόν η επανάσταση από νέα παιδιά, μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου, ε, φοιτητές πανεπιστημίου, που είπαν έχουμε βαρεθεί τον και Θέλουμε τη δημοκρατία, θέλουμε ελευθερίες, θέλουμε να ζούμε σε ένα καλύτερο κόσμο. Τώρα που θυμάμαι ξανά εκείνες τις εποχές, ε, όπως και άλλοι 50χρονοι νέοι, ερχόμαστε και δίνουμε τη μαρτυρία μας πώς αξιοποιήσαμε, πώς χρησιμοποιήσαμε αυτά τα 30 χρόνια ελευθερίας και δημοκρατικής κοινωνίας. Οι περισσότερες ιστορίες είναι πολύ πετυχημένες και πολύ ευτυχισμένες και ξέρω τι σημαίνει όταν αγωνίζονται οι νέοι, αγωνίζονται για ένα καλύτερο μέλλον και όσο μπορώ από τη νέα μου θέση θα σας βοηθήσω και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η ΑΚΡΑΤ έφτασε στις κάτω χώρες ε, εδώ και αρκετά χρόνια από το Ιρακινό Κουρδιστάν και θα μας διηγηθεί την ιστορία της όπως έκανε και η κυρία Γιώροβα. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες, Σακράτ. Έχεις το λόγο. Ε, σκέφτηκα για πολλή ώρα τι να πω και τι να μην πω σε αυτό το χώρο, σε αυτή την πολύ όμορφη και πολύ σημαντική ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού. Σκέφτηκα να μιλήσω για την παιδική μου ηλικία που μου τη στέρισαν κατά την παραμονή μου στην, ε, στις κάτω χώρες αφού έφυγα από τη χώρα μου για να γλιτώσω να μιλήσω για τις μετακομίσεις που κάναμε πέντε φορές μέσα σε ένα χρόνο, δηλαδή να χρειάστηκε να αφήσω το σπίτι μου, τους φίλους μου, τη γειτονιά μου, την ασφάλειά μου, πέντε φορές μέσα σε ένα χρόνο. Θα μπορούσα επίση να σα μιλήσω για το γεγονό ότι χρειάστηκε για δύο χρόνια να πηγαίνω ερχόμαστε στα δικαστήρια για να πάρουμε μια ιατρική καρέκλα μπάνιου για την μικρή μου αδερφή που έχει σωματική και ψυχική αναπηρία. Ή να σας μιλήσω για το γεγονός ότι έπρεπε να συγκατοικώ με έξι μέλη της οικογένειάς μου σε ένα δωμάτιο και για την έλλειψη ιδιωτικότητας που βίωσα. Για το γεγονός ότι παιδιά και έφηβοι χωρίς χαρτιά δεν έχουν το δικαίωμα ε, για πλήρη παιδεία, ε, για πλήρη εκπαίδευση, όταν φτάνουν στα 18 και επιπλέον δεν έχουν την ικανότητα να συναποφασίζουν για θέματα που αφορούν αυτά τα παιδιά και αυτούς τους εφήβους άμεσα. Υπάρχουν τόσα πολλά που θα ήθελα να σας πω, αλλά αυτό που θα ήθελα κυρίως να σας πω είναι αφήστε τα παιδιά να είναι παιδιά. Σας ευχαριστώ. Ονομάζομαι Αχράτ Σελεβάνη. Ευχαριστούμε, Χράτ. Και τώρα λόγω στον κύριο Φλάχερτη. Ήρθε η σειρά σας, κύριο Φλάχερτη. Καλώς ήρθατε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε με την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή τη διάσκεψη ψηλού επίπεδου. Ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΑΧΡΑΤ για τα βαρισίμαντα λόγια που μας απευθύνε. Είναι η πρώτη νεαρή που μίλησε και άξιζε η ώρα που περίμενα για να ακούσω αυτά τα σπουδαία λόγια της Αχράτης. Ευχαριστώ θερμά. Οφείλω να ομολογήσω ότι σήμερα νιώθω αρκετά γερασμένος όχι γιατί έχουμε τόσο νέους, τόσους πολλούς νέους στην αίθουσα, γιατί θυμάμαι ακόμη με σαφήνεια την ημέρα του 1989 όταν υιοθετήσαμε τη σύμβαση. Βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη και θυμάμαι όλες τις εφημερίδες που είχαν πρωτοσέλιδα της, την είδηση για την κύρωση αυτής της ηθίκης ε, με συμμετοχή ε, χωρών από όλες τις γωνιές του κόσμου. Και θυμάμαι πόσο συνεργασμένοι ήμασταν για το περιεχόμενο της ηθίκης, γιατί ήταν και τότε αλλά και τώρα η συνθήκη αυτή είναι ριζοσπαστικό εργαλείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλούσε για το παιδί ως ανθρώπινο πλάσμα, ως ανθρώπινο όν που δεν ε, χρήζει μόνο προστασίας αλλά ε, θα πρέπει να έχει και το δικαίωμα να εκφέρει τη γνώμη του και είναι βασικός φορέας ε, και κάτοχος δικαιωμάτων για κάθε δράση που το επηρεάζει. Ακόμη και με τον ενθουσιασμό του 1989 δύσκολο θα ήταν να προβλέψουμε τι ρηξικέλευθες αλλαγές θα έφερνε η σύμβαση αυτή την 30 ετία που ακολούθησε και έχουμε τόσα παραδείγματα για το πώς άλλαξε το κόσμο. Κοιτάξτε UNICEF. Μεταμόρφωσε τη UNICEF. Τότε η UNICEF ήταν ε, ο ισχυρότερος παράγοντας του ανθρωπιστικού έργου στα Ηνωμένα Έθνη. Και η UNICEF ήταν η ατμομηχανή για την ανάπτυξη μιας προσέγγισης που θα δράζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και έτσι οδηγηθήκαμε στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Και σε ό,τι αφορά το εθνικό επίπεδο, ε, έχουμε συνηγόρου των δικαιωμάτων του παιδιού σε τόσα πολλά χρόνια. Έχουμε ε, σχέδια δράση για τα δικαιώματα του παιδιού σε τόσα πολλά μέρη του κόσμου. Χάρη στη σύμβαση αυτή. Η σύμβαση αποτέλεσε τη βάση για πολύ σημαντικά εθνικά μέτρα και πρωτοπορία εθνική σε τέτοια μέτρα σε πολλέ χώρε του κόσμου. Και χαίρομαι που ε, είμαι εδώ με την πρόεδρο Κολέρα Πρέκα που ήταν πολύ σημαντική ηγετική μορφή στα θέματα αυτά. Και όπως είπε και η Επίτροπος ε, Γιώροβα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού πυροδότησε τεράστιο αριθμό νομοθετικών διατάξεων που πραγματικά έχουν επιφέρει μεγάλες αλλαγές. Μία σημαντική νομοθετική αλλαγή ήταν ε, ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων που είναι το εργαλείο θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 24 του χάρτη αυτού εμπνέεται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Και η εγγύηση για τα δικαιώματα του παιδιού του χάρτη θεμελιών δικαιωμάτων δεν θα ήταν τόσο σημαντική και τόσο ευρεία αν δεν ακολουθούσε την έμπνευση της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού. Και έχουμε πολλούς λόγους για εορτασμό σήμερα. Αλλά Άκουσα στην εναρκτήρια τελετή και άκουσε και από την ομιλία της Επιτρόπου Γιώροβα και από αυτά που μας είπε η Ακράτ ότι έχουμε ακόμη μακρύτερα δρόμο μπροστά μας. Οπότε δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μα ούτε να αδρανούμε. Εγώ θα επικεντρωθώ σε τρει τομεί που σε μεγάλο βαθμό εμ, συμπίπτουν με αυτά που μα είπε η κυρία Γιώροβα. Και ο πρώτο τομέα είναι η μετανάστευση. Η κατάσταση των παιδιών ε, ε, μεταναστών είναι ιδιαίτερα προβληματική και ανησυχητική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από δύο εβδομάδες είχα επισκεφθεί τον καταβλισμό της Μόριας και το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στο νησί της Λέσβου στην Ελλάδα. Εκεί διαπιστώνουμε το εύρος των προκλήσεων, ε, ειδικά για τα παιδιά. Τη μέρα που πήγα στη Μόρια είχαμε περίπου χίλια συνόδευτα παιδιά, χωρίς κηδεμόνες, χωρίς επιμελητές, χωρίς ε, γονείς. Και μόνο 300 από τα χίλια αυτά παιδιά βρισκόταν σε ένα ασφαλές μέρος για παιδιά. Τα υπόλοιπα 700 παιδιά ήταν ασυνόδευτα στον καταβλισμό χωρίς ειδική προστασία. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Θυμάμαι ένα παιδί ε, τότε, τη μέρα που φεύγαμε ε, από την ασφαλή ζώνη για τα παιδιά, ήταν ένα 12χρονο περίπου αγόρι και είδα ότι στο μπράτσο του είχε ένα πολύ μεγάλο τατουάζ και αυτό που με ενόχλησε ήταν η εικόνα του τατουάζ. Ήταν ένα όπλο Καλάσνικοφ. Ρώτησε λοιπόν το παιδί, γιατί, γιατί αυτό το τατουάζ, γιατί έχεις το τατουάζ με το Καλάσνικοφ και μου απάντησε γιατί μου υπενθυμίζει ότι στον κόσμο αυτό θα πρέπει κανείς αν θέλει να επιβιώσει πρέπει να αγωνιστεί. Κανένα παιδί σε αυτήν την ηλικία δεν θα πρέπει να λέει κάτι τόσο σοκαριστικό. Όπως είπα λοιπόν το θέμα των hot spot και των κέντρων υποδοχής για τους ε, μετανάστες και τους πρόσφυγες είναι πολύ ενισχυτικό. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι η ανάγκη για καλύτερη ε, δουλειά που θα πρέπει να κάνουμε στην κοινωνική ένταξη των παιδιών. Από τη στιγμή που περάσουμε τις πρώτες διαδικασίες της υποδοχής και ξεκινήσουμε στο στάδιο της ένταξης, εκεί θα πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση. Χθε, ο Οργανισμό Ανθρωπίνων Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δημοσίευσε μία έκθεση για την εμπειρία των νέων που έφτασαν στην Ευρώπη το 2015 και το 2016. Και σίγουρα υπάρχουν μερικέ καλέ πρακτικέ, αλλά δυστυχώ είχαμε πολύ περισσότερε ανησυχητικέ εξελίξει σε πολλά σημεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και περνάμε από τη μετανάστευση στο θέμα τη φτώχεια. Και εδώ θα πρέπει να διατηρήσουμε την εξάλληψη της φτώχειας, της παιδικής φτώχειας ως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1 τέταρτο του συνόλου των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν σε φτωχά νοικοκυριά, σε φτωχές οικογένειες. Δηλαδή 25 εκατομμύρια παιδιά ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Και μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι από τις πλουσιότερες και πιο εύπορες γωνιές του κόσμου. Και αν ε, ξεπεράσουμε τα γενικά νούμερα και επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες ομάδες, η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική. Όπως λοιπόν και η κυρία Γιώροβα, εγώ θα ήθελα να σταθώ στην κατάσταση των παιδιών Ρωμά. 6 εκατομμύρια είναι τα μέλη των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα σας δώσω ένα μόνο αριθμητικό στοιχείο. 41% δηλαδή τα μισά περίπου παιδιά Ρωμά μένουν σε οικογένειες ή σε νοικοκυριά όπου ένα τουλάχιστον μέλος του νοικοκυριού πηγαίνει να κοιμηθεί νηστικό. 41% σχεδόν τα μισά παιδιά Ρωμά. Αυτό είναι σοκαριστικό. Γιατί αν θέσουμε την ίδια ερώτηση στο ευρύ κοινό, στην υπόλοιπη κοινωνία, αν ρωτήσουμε λοιπόν το γενικό πληθυσμό πόσα παιδιά μένουν οικογένειες οικογένειε που ένα πάει να κοιμηθεί νηστικό είναι 8% σε σχέση με το 41% που είναι το ποσοστό στην κοινότητα Ρωμά και 8% το ποσοστό στο γενικό πληθυσμό. Και τρίτο και ε, πολύ ανησυχητικό θέμα είναι το ζήτημα των παιδιών στο δικαιικό σύστημα, στο δικαστικό σύστημα. Τα παιδιά ως μάρτυρες, ε, ως ε, αντικείμενα προσοχής στις διαδικασίες διαζυγίου ή στις διαδικασίες υιοθεσίας και σε όλες τις πτυχέ του δικαστικού συστήματος. Θέλουμε μια δικαιοσύνη που θα είναι φιλική προς τα παιδιά. Δυστυχώς όμως ο οργανισμός μας επανειλημμένος αποκάλυψε πολλές περιπτώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε δυστυχώς εχθρική προς το, προς το παιδί δικαιοσύνη και απόλυτη έλλειψη προσοχής και φροντίδας για τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν τα παιδιά και μπορεί πραγματικά να τραυματίσουμε πολύ τα παιδιά από απερισκεψία στη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Και έρχομαι στο τελευταίο σκέλος της ομιλίας μου ε, που περνάει από τις ανησυχίες της δράσης. Εμείς στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων εξετάζουμε συγκεκριμένες δράσεις. Για παράδειγμα, σας μίλησα πρώτα για την κατάσταση των παιδιών μεταναστών. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την προστασία των παιδιών και δεν μπορούμε να το κάνουμε αν δεν επικεντρωθούμε στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης αλλά ε, και στη μεταγενέστερη φάση, τη φάση της κοινωνικής ένταξης. Θα πρέπει η ένταξη να λάβει υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κρατη και πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε, όχι μόνο με ανταλλαγή βέλτιση των πρακτικών. Επίσης, παιδική φτώχεια. Μία και μόνο σύσταση έχω. Το σύστημα εγγύησης ε, για τα παιδιά είναι μια καταπληκτική ιδέα που αναπτυχθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι δύσκολο βέβαια να υλοποιηθεί. Θα πρέπει να συνεργαστούν τα τρία θεσμικά όργανα, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πραγματικά θα αλλάξει την κατάσταση για τα παιδιά. Επίση, τα παιδιά στο δικαστικό σύστημα. Θα πρέπει να βελτιώσουμε την εφαρμογή τη υπάρχουσα νομοθεσία και να επενδύσουμε σε κατάρτιση και πόρου για να υλοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές. Σήμερα είναι μια πανέμορφη μέρα γιατί εορτάζουμε και εδώ και παγκοσμίω αυτή την Διεθνή Σύμβαση και γι' αυτό θα πρέπει ε, να φροντίσουμε ότι, ώστε την επόμενη τριακονταετία οι αλλαγές να είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εσείς οι νέοι ε, μεταξύ των νέων ε, υπάρχουν νέοι που είναι δραστήριοι. Στο πρωτόκολλο 3 για ε, το πρωτόκολλο των παιδιών δίνει την ευκαιρία ε, να ε, το αξιοποιήσουν τα παιδιά και το έχει κάνει η Ράινα και κάποιοι άλλοι νέοι ε, για να διεκδικήσει αυτά τα δικαιώματα. Έχει το λόγο Ράινα. Ευχαριστώ πολύ. Ήρθα εδώ σήμερα γιατί η κλιματική κρίση είναι η πιο μεγάλη απειλή στα δικαιώματα των παιδιών. Το δικαίωμα που μου έχουν τάξει και εμένα και σε όλα τα παιδιά πριν από 30 χρόνια και σε όλα τα παιδιά αυτού του κόσμου. Η κλιματική κρίση είναι η μεγαλύτερη απειλή. Όχι απλώς για το δικό μου μέλλον και για το δικό μου σπίτι, αλλά ήδη καταστρέφει εκατομμύρια ζωές αυτή τη στιγμή που μιλάω. Migration. Η μετανάστευση, η πόλεμη και η φτώχεια στο μέλλον θα χειροτερέψουν ε, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης. Ε, ε, εδώ βλέπουμε ο κόσμος να συνεχίζει να επενδύει στα ορυκτά καύσιμα ενώ τα παιδιά πεθαίνουν καθημερινά και συνεχίζουν να πεθαίνουν. Όπως είπα, η κλιματική κρίση θα δημιουργήσει εκατομμύρια προσφύγων και για την Ευρώπη ή τη Γερμανία τουλάχιστον Μπορώ να πω ότι δεν μπορούμε να δώσουμε ασφαλή στέγη στους ανθρώπους αυτούς. Τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία ήρθαν λίγα εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν μπόρεσαν να τους στεγάσουν με ασφάλεια. Και στο μέλλον πώς θα το κάνουμε αν έχουμε 500 εκατομμύρια να δώσουμε στον κόσμο αυτό στέγη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα δεν θέλω να σας κάνω διδάγματα, αλλά το σπίτι μου αλλάζει και η κυβέρνησή μου αδρανεί και αυτό με τρομάζει. Στη Γερμανία φέτος ζήσαμε το χειρότερο καλοκαίρι, το πιο ζεστό όλων των εποχών. Και ε, όχι μόνο το καλοκαίρι και ο χειμώνας ε, είναι πιο θερμός. Στο Αμβούργο δεν χιονίζει πια. Δεν βλέπουμε χιόνι. Ε, έχουμε πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Κάναμε λοιπόν μια αναφορά και με τους φίλους μου στα νησιά Μάρσαλ. Και εγώ πραγματικά είμαι εξαιρετικά προνομιούχα αν συγκρίνω τη δική μου ζωή με τη δική τους. Οι άνθρωποι αυτοί χάνουν τα σπίτια τους όπως και πολλοί άλλοι νησιώτες. Την ώρα που μιλάμε. Αυτό θέλω να τονίσω. Και δεν χάνουν μόνο τα σπίτια τους, τους φίλους τους, τα αδέλφια τους, τις οικογένειές τους. Και εμείς καθόμαστε εδώ και συζητάμε. Ζούνε τους χειρότερους εφιάλτες λόγω της δικής μας γελίας κατανάλωσης. Οι άνθρωποι αυτοί που ζουν με τρόπο απλό και παραδοσιακό πλήττονται περισσότερο και πιο σφοδρά από την κλιματική κρίση. Και αυτή τη στιγμή η Γερμανία και η Κάρβουνο. Αλλά και εγώ ζω στη βολή μου. Αυτά τα πράγματα μου ακούγονται άδικα. Η Γερμανία τέλος έχει τεράστιο οικολογικό αντίκτυπο. Εμείς επενδύουμε σε ε, ορυκτά καύσιμα και οι άνθρωποι αυτοί χάνουν τα σπίτια τους. Εμείς ε, τους προκαλούμε το φόβο και τα δεινά. Και αυτοί οι άνθρωποι, φίλοι μου, ε, φοβούνται κάθε μέρα ο τρόπος με τον οποίο ζούμε εμείς στη Γερμανία, οι περισσότεροι και αλλού στην Ευρώπη, εντείνει την κλιματική αλλαγή και τα προβλήματα. Και ως παιδιά μαθαίνουμε να νοιαζόμαστε για τους άλλους, να βοηθάμε εκείνους που μας χρειάζονται. Αλλά φοβάμαι ότι οι ηγέτες, οι παγκόσμιοι και πολλοί ενηλικοί καθώς ενηλικιώνονται, αλλά αυτά τα ξεχνάνε. Θα πρέπει οι ηγέτες μας λοιπόν οι παγκόσμιοι να σταματήσουν να βάζουν πρώτα το κέρδος και μετά τον άνθρωπο και να μας δώσουν τα δικαιώματα που μας έταξαν. Το μόνο που ζητώ είναι βασικά θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιώματα του παιδιού. Δεν ζητώ λαγούς με πετραχίλια. Και είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Και θα πρέπει τώρα να το αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι δικαίωμά μου και δικαίωμα κάθε παιδιού να έχει μέλλον και μια ασφαλή στέγη. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τις διαφορές μας και να συνεργαστούμε όχι μόνο στην πολιτική αλλά στις πόλεις, στους δήμους και κοινότητες. Και μια που πρόκειται για το δικό μας μέλλον θα πρέπει να είμαστε και τμήμα της συζήτησης. Θα πρέπει να συμμετέχουμε στις αποφάσεις και όχι να αγωνιζόμαστε για να επιβιώσουμε και να ε, κάνουμε σκάση αρχείο για να διαδηλώνουμε. Μας έχουν υποσχεθεί προστασία αλλά δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους. Θα πρέπει να συμμετέχουμε στη διαδικασία. Ειλικρινά σας λέω ότι έχω μπουχτίσει να ζητάω τα δικαιώματά μου όταν οι παγκόσμιοι ηγέτες υποκρίνονται ακόμα ότι δεν ακούν τη φωνή μου. Δεν θα σας αφήσουμε το χώρο να περιμένετε παίρνουμε την ευκαιρία και δρούμε, τουλάχιστον για παράδειγμα κάθε Παρασκευή. Ασχοληθείτε με αυτή την κλιματική κρίση και καταλάβετε ότι είναι κρίση και έκτακτη ανάγκη, γιατί εγώ θέλω να επιβεώσω και να έχω και μέλλον. Ευχαριστώ. Bien. Muchas gracias, Reina. Σιώδα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Σιόντα έχει τώρα εμπειρία από τα τοπικά συμβούλια γιατί για τα παιδιά ασχολούνται με αυτά σε επίπεδο και με τα δικαιώματα τους. Ευχαριστούμε που ήρθες, έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Σίντι. Είμαι 14 και είμαι από την I'm a member of the Eurochild Council. Είμαι μέλος του Συμβουλίου Παιδιών της Eurochild που είναι μια οργάνωση που προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά που θα αναπτύσσονται θα μεγαλώνουν χαρούμενα με υγεία και με σεβασμό από πλευράς της κοινωνίας ε, με σεβασμό στους άνθρωποι ως φυσικά πρόσωπα και έχω με άλλους 11 και εκπροσωπούμε διάφορους ε, άλλου φορεί ε, για τοπικέ δραστηριότητε και σήμερα μιλώ εκ μέρου αυτού του συμβουλίου του Eurochild. Γιατί είμαστε εδώ, Γιατί πάρα πολλοί από του πρωθυπουργού μα και τη δική μου χώρα έχουν έρθει σε αυτό το ίδιο ημικύκλιο και έχουν ε, πει το πώ βλέπουν το μέλλον τη Ευρώπη, το όραμά του, αλλά κανένα δεν επηρεάζεται περισσότερο από τις εξελίξεις του μέλλοντος από τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ. Γι' αυτό ήρθα να σας πω ότι γίνεται με τα παιδιά σαν και εμένα. Ε, τι Ευρώπη θέλουμε. Και σήμερα επίσης μιλώ για λογαριασμό των 20.000 παιδιών που ε, συμμετέσχουν στην έρευνα που ε, κάναμε ε, Europe Kids Want ε, σήμερα σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια ο κόσμος αναγνώρισε τα δικαιώματά μας των παιδιών και μας δίνει ε, δικαιώματα που θα έπρεπε να έχουν όλοι οι άνθρωποι ε, στην γη. Αυτό μπορεί να φαίνεται πάρα πολύ χαριτωμένο αλλά δεν έχει γίνει ακόμα πραγματικότητα γιατί οι παιδιά ε, σκοτώνονται, βιάζονται, πρέπει να δουλεύουν σε λίγο πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν είναι σωστό, θα έπρεπε να τα φροντίζουν τα παιδιά, θα τα στέλνουν στο σχολείο για να έχουν ασφάλεια. Και ε, ε, ρωτήσαμε πέρσι τα παιδιά στην Ευρώπη τι Ευρώπη θέλουν από Σερβία, Σλοβακία ε, μέχρι Γαλλία και Φιλανδία όλα τα παιδιά ανησυχούσαν ως αυτό το μέλλον της Ευρώπης και ήρθαμε εδώ για να σας ακριβώς εκφράσουμε αυτές τις ανησυχίες πρόκειται για 23 εκατομμύρια παιδιά δηλαδή ένα στα τέσσερα που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας το Child Poverty ασχολείται με όλα αυτά τα προβλήματα των παιδιών, με τους νέους επίσης για το πώς θα αποκτήσουν δεξιότητες, πώς θα βοηθήσει το Child Poverty ε, για τα προβλήματα, τα προβλήματα συμπεριφοράς κοινωνικά ε, και συναισθηματικά Με την ανεργία ε, με τα άστεγα παιδιά και με θέματα πνευματικής ε, συναισθηματικής υγείας και επίσης έχουμε παιδιά κάθε ηλικία που ανησυχούν για το bullying μέσω του ίντερνετ και πάρα πολύ έχουμε προσπαθήσει να χρησιμοποιήσουμε τους κατάλληλους διάβλους ούτως ώστε το ίντερνετ να είναι ασφαλές ναι, υποφέρουν τα παιδιά όμως υπάρχει ελπίδα αλλαγής, υπάρχει το κατάλληλο κλίμα και αυτή είναι οι προτεραιότητές μας. Έχουμε παλέψει στο μέτωπο της φτώχειας για τα παιδιά, έχουμε αυτή την έρευνα, στείλουμε στα σχολεία να ακούσουμε τη γνώμη των παιδιών και επίσης προσπαθούμε όσον αφορά το περιβάλλον και επίσης ε, την εγκληματικότητα. Αλλά έχουμε και κάποια προβλήματα γιατί όταν προτάσουν τα δικαιώματά μας πάρα πολλοί μας είπαν να σιωπήσουμε και να κάτσουμε στη θέση μας. Μα λένε ότι δεν είναι σημαντική η γνώμη μας γιατί είμαστε πάρα πολύ νέοι. μα είπαν ότι δεν έχουμε το δικαίωμα του να ακούγεται η φωνή μα. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν ισχύει. Θεωρούμε ότι όλα αυτά ε, θα έχουν επιπτώσεις, ε, όλα αυτά θα είναι κίνητρα για να φέρουμε την ε, αλλαγή. Και βέβαια δεν περιμένουμε να μας τα φέρουν όλα έτοιμα. Πιστεύουμε ότι με τις γνώμες μας μπορούμε να αλλάξουμε την μοίρα της Ευρώπης. Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε υποπροϊόντα. Είμαστε το παρόν 20% του πληθυσμού της Ευρώπης, είμαστε το 100% του μέλλοντο που οικοδομείται. Οπότε δεν είμαστε εδώ μόνο για να επαναστατήσουμε, για να, για να, ούτε για να σας διαβάσουμε στατιστικές από το χαρτί αυτό, αλλά ήρθαμε εδώ για να αναλάβουμε δράση γιατί θέλουμε να υπάρχει μια διαρκή και πραγματική αλλαγή. Τι χρειαζόμαστε από εσά, Εσεί διαμορφώνεται τι αποφάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσεί χαράζετε πολιτικέ και θεσπίζετε κανόνε και ξέρουμε ότι έχετε την ευφυα και την εμπειρία να φτιάξετε ένα καλύτερο μέλλον για μα. Και θέλουμε αυτό να το κάνετε με την άμεση συμμετοχή μα, εμπλοκή μα. Θέλουμε καλύτερου κανόνε από του ενήλικου, ούτω ώστε να προστατεύουν τα δικαιώματά μα και να εξασφαλίσετε ότι θα υπάρξει παιδεία στη βάση των δικαιωμάτων. Και θέλουμε να κάτσουμε στο τραπέζι, να συζητήσουμε του κανόνε μαζί σα, εσεί που λαμβάνετε τι αποφάσει, να ακούσετε, να λάβετε υπόψη τι γνώμες μας το καλοκαίρι. Έγινε ε, μια αναφορά, μια, ένα, ψήφισμα για να ζητηθεί να θεσμοθετηθεί Ευρωπαίος Επίτροπος για τα παιδιά. Αυτό θα ε, δεν θα πρέπει να χρειάζεται να γίνει. Γιατί θα έπρεπε ότι αφού είναι πρωτοπόρα η Ευρώπη στον κόσμο, στα δικαιώματα θα έπρεπε να έχει τέτοιον επίτροπο και δικαιώματα των παιδιών στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία. Επίση, είχαμε κάποια διακήρυξη από παιδιά ε, και πρέπει να συνεργαστούμε και να συνεργαστούμε για να εξασφαλιστεί ε, η χαρά, η υγεία για τα παιδιά, η ανεμπόδιστη ανάπτυξη, ούτω ώστε να μην χρειάζεται να δώσουμε ένωση για τα δικαιώματα. Και σύμφωνα με την σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα, οι απόψεις μας λαμβάνονται υπόψη και θα πρέπει τα συμφέροντά μας να είναι η κορυφαία προτεραιότητα. Θα πρέπει για κάθε ψηφοφορία να σκέφτεστε δύο φορές κατά πόσο η σχετική απόφαση θα βοηθήσει τα παιδιά. Να εξασφαλίσετε ότι μπροστά μας το μέλλον θα είναι ρόδινο για να είμαστε προετοιμασμένοι, εκπαιδευμένοι, ούτως ώστε να ωφεληθεί και ο κόσμος και εμείς. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα καινοτόμο με απόδοση ευθυνών χωρίς αποκλεισμούς. Θέλουμε να υπάρξει ε, επένδυση εκεί που χρειάζεται, δηλαδή υγεία, ε, παιδεία, διατροφή, κοινωνική πρόνοια, ε, ιατρική κάλυψη, όλα αυτά θα πρέπει να καλύπτονται από εσωτερικέ και εξωτερικέ πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε αλληλεγγύη με τα παιδιά σε όλο τον κόσμο. Έκλεισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει κατεπίγοντα μέτρα να προστατευτεί το περιβάλλον. Εμεί θα πρέπει αύριο να ζήσουμε και να υποστούμε τι συνέπειε των σημερινών πολιτικών αποφάσεων. Τέλο, θέλουμε εσεί να παίρνετε τι αποφάσει όλα αυτά να τα πάρετε σοβαρά, να μην τα υποτιμάτε δεν ε, είμαστε αντιρρησίες, δεν είμαστε στασιαστές απλώς μας καίνε τα δικαιώματα της γενιάς μας πρέπει να αλλάξουμε, μπορούμε να αλλάξουμε το πρόσωπο της ε, υπήρου μας Una de ε, κάτι που συμβαίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα και αν δεν τηρήσουμε όλοι αυστηρά το χρόνο μας θα στερήσουμε τη δυνατότητα από τους επόμενους ομιλητές ε, να λάβουν το λόγο. Η κυρία Πρέκα θα μας πει για το πώς ασκούνται τα δικαιώματα αυτά στη δική μας περιοχή. Θα είναι πολύ δύσκολο να ε, παίρνει κανείς το λόγο μετά από αυτά τα καταπληκτικά παιδιά που μας εξήγησαν τόσο καλά την κατάσταση και τις προσδοκίες τους, που είναι κοινέ με αυτές άλλων παιδιών. Όταν η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ε, ήταν αναφυσβήτητα ο φάρος για τα δικαιώματα των παιδιών παγκοσμίω, διαμόρφωσε την προσέγγισή μας για τα δικαιώματα του παιδιού. Επίσης, ε, μας έδωσε ένα πλαίσιο όπου πολιτικές συναφεί με τα δικαιώματα των παιδιών θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και διεθνές επίπεδο. Από πρακτική άποψη, η διεθνής αυτή σύμβαση και τα πρωτόκολλά τη βοήθησαν ε, στο να βελτιωθεί η κατάσταση εκατομμυρίων παιδιών. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων και η διαδικασία της, του σχεδιασμού της οικίας νομοθεσίας και των οικιών πολιτικών ε, συνεχίζει να ε, εξωθείται χάρη στην διεθνή αυτή σύμβαση. Βέβαια δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι το έργο μας για τα δικαιώματα του παιδιού έχει ολοκληρωθεί. Στο μέτρο που η Ευρώπη και ο κόσμος ε, ε, βαδίζουν προς τη νέα αυτή χιλιετία, νέες προκλήσεις αναδύονται και μερικές φορές οι παλιές προκλήσεις επανέρχονται και μας τυχιώνουν. Το, δημοκρατικό, το δημογραφικό τοπίο της Ευρώπης αλλάζει. Οι οικονομίες επεκτείνονται και συρρυκνώνονται. Σκληροπυρηνική πολιτική αντικαθιστούν πιο μετριοπαθείς. Οι εξελίξεις είναι ορατέ στις γειτονικέ μας περιοχέ και οι προκλήσεις για τα παιδιά και τι κοινωνίε μα εξελίσσονται. Τα ευάλωτα μέλη των κοινωνιών μα είναι αυτά που πλήττονται περισσότερο από όλε αυτέ τι αλλαγέ. Ε, αυτοί που δεν έχουν εξουσία, δεν έχουν φωνή, μερικέ φορέ δεν έχουν καν ψήφο. Και τα παιδιά εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Και πέτοι όπω αυτή μας υπενθυμίζουν τη σημασία που έχει η συνέχιση του έργου μας προκειμένου να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των παιδιών. Γιατί πολύ δρόμο έχουμε ακόμη μπροστά μας. Πολύ έργο θα πρέπει να επιτελεστεί ώστε κάθε παιδί να μπορεί πραγματικά να επιβιώσει και να ευημερήσει. Δυστυχώς έχουμε πολλά εμπόδια που θα πρέπει να υπερκεράσουμε στην προσπάθεια αυτή. Εγώ θα επικεντρωθώ σε τρία μόνο βασικά εμπόδια, δηλαδή στη φτώχεια, τη μετανάστευση και την αναπηρία ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ακούσαμε, βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες η παιδική φτώχεια φτάνει σε ποσοστό άνω των 40%. Οι στατιστικές λοιπόν σίγουρα δεν προμηνύουν κάτι καλό. Γιατί όχι μόνο αυτά τα παιδιά δεν πρόκειται ουδέποτε να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους, αλλά γνωρίζουμε ότι παιδιά από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος ε, κατά πάσα πιθανότητα θα παρατήσουν και το σχολείο. Επίσης γνωρίζουμε ότι παιδιά από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος ε, έχουν τριπλάσιο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας ή ψυχικής υγείας. Επίσης, ε, υποφέρουν καθόλου τη διάρκεια της ζωής τους και πολύ συχνά παρατάνουν νωρί στο σχολείο. Επίσης ε, έχουν ε, μεγάλες προκλήσεις ε, και προβλήματα υγείας ή ψυχικής υγείας και είναι διαβίου σε μειονεκτική θέση σε σχέση με παιδιά από εύπορε οικογένειε. Και το σενάριο τη πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Γιατί μελέτε επισημαίνουν στενούς δεσμούς μεταξύ της πρόορης εγκατάλειψης ε, του σχολείου και μεγάλων πτυχών της ευημερίας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Θα πρέπει λοιπόν να διασπάσουμε αυτόν τον κύκλο. Κάτι που απαιτεί τεράστιε προσπάθειε. Και όσο περισσότερο χρόνο περάσει, τόσο μεγαλύτερε προσπάθειε θα πρέπει να κάνουμε για να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ των ευπόρων και των απόρων, που όλο και μεγαλώνει. Στο μεταξύ, το πεπρωμένο αυτών των παιδιών θα έχει προκαθοριστεί, γιατί τα παιδιά που γεννιούνται στη φτώχεια κατά πάσα πιθανότητα μεγαλώνουν και φτωχά, φτωχά και πολύ πιθανό μεταβιβάζουν αυτή την κατάσταση και στην επόμενη γενιά. Θα ήθελα τώρα να πω λίγα λόγια για τα παιδιά στη μετανάστευση. Πάνω από 30.000 ε, παιδιά μεταναστών και προσφυγόπουλα ε, αγνοούνται στην Ευρώπη μεταξύ του 2014 και του 2017. Αυτά τα νούμερα είναι σοκαριστικά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε παιδί βρίσκεται μια θλιβερή ιστορία απόγνωσης. Τα παιδιά αυτά αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις αιστείες τους και μετά περνά τα πάνδυνα ε, κατά τη διάρκεια χρονοβόρων και επικίνδυνων ταξιδιών και τελικά καταλήγουν σε χώρες που είναι απροετοίμαστες και πολύ συχνά και απρόθυμες να αναλάβουν την ευθύνη της προστασίας τους και να εξασφαλίσουν το σεβασμό των στοιχειωδών και θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Και μάλιστα η φετινή έκδοση της διάσκεψης ε, χαμένη στη μετανάστευση που έγινε στην Μάλτα εξετάζει αυτό το θέμα της εξαφάνισης παιδιών στην Ευρώπη. Γιατί έγινε η ανάλυση της κατάστασης και επιβλήθησαν πολλές συστάσεις για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανθρώπινη τραγωδία που σημαίνει και εδώ και αλλού. Και ένα άλλο σημαντικό έγγραφο που εκθέτει αυτή την κατάσταση και υποβάλλει πολύ σημαντικές στάσεις είναι το άγραφο της Eurochild για το «Σώστε τα παιδιά». Επίσης, ε, θα πρέπει να αλλάξει το αφήγημα γύρω από τη μετανάστευση και ιδιαίτερα των παιδιών μεταναστών. Θα πρέπει να, μεταμορφ... να μετατρέψουμε αυτό το αφήγημα και να εξασφαλίσουμε συνέστηση για τα παιδιά στήριγμα, βοήθεια και χειραφέτηση. Επίσης θα πρέπει να έχουμε πολιτικές διαχείρισης τη μετανάστευσης για να υλοποιήσουμε πραγματικά τα δικαιώματα των παιδιών και να ε, εξασφαλίσουμε ε, την ε, μέρημνα του υπέρτερου συμφέροντος του παιδιού. Η UNICEF υπολόγισε επίσης ότι τα παιδιά με αναπηρίες έχουν τριπλάσια ή τετραπλάσια πιθανότητα να γίνουν θύματα σωματικής και σεξουαλικής βίας ή παραμέλησης από ότι τα μέλη παιδιά. Τα παιδιά με αναπηρίες έχουν καθημερινά εμπόδια στη ζωή τους και στην ευημερία τους. Επίσης φέρουν το στίγμα και τη διακριτική μεταχείριση. Και μερικές φορές ο αγώνας τους είναι αφανής. Θα ήθελα να σας πω μια ιστορία για το εμπόδιο που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρία στην Ευρώπη. Μια οργάνωση στην οποία προεδρεύω στη Μάλτα έχει ένα συμβούλιο παιδιών και ένα συμβούλιο νέων. Πριν από λίγα χρόνια Μερικά από τα παιδιά μας προσκλήθηκαν να συμμετέχουν σε μια συνεδρίαση εδώ στις Βρυξέλλες. Ένα παιδί που ε, ήταν ανάπηρο και χρειαζόταν ε, αναπηρική πολυθρόνα συμμετείχε σε αυτή την αντιπροσωπεία. Και το ταξίδι του ήταν γεμάτο προσκόμματα και εμπόδια, δυσκολίες που δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζει κανένα παιδί. Και το πρώτο πρόβλημα το είχε πριν καν ε, ξεκινήσει η πτήση του, γιατί έπρεπε να απενεργοποιήσουν την μπαταρία της ε, αναπηρικής πολυθρόνας, κάτι που καθυστέρησε την πτήση και από τη στιγμή που προσγειώθηκε επίσης ε, δεν μπορούσε να μεταφερθεί ε, στο ξενοδοχείο του. Και μετά από πολλά τηλεφωνήματα τελικά βρήκαμε ταξί, αλλά συνεχίστηκε μέχρι το ξενοδοχείο το πρόβλημα. Μάλιστα το ξενοδοχείο είχε επιβεβαιώσει ότι ήταν κατάλληλα εξοπλισμένο για αναπήρους, κάτι όμως που δεν ίσχυε για το λουτρό. Οπότε δημιουργήθηκαν ακόμη μεγαλύτερε δυσκολίε για το παιδί. Συνεχίστηκαν τα προβλήματα ε, στα εστιατόρια που πήγε και στη μετακίνηση του από το ένα μέρος στο άλλο. Και ε, η τραγική ηρωνία ήταν ότι το αντικείμενο τη συνεδρίαση ήταν η προστασία των θεμελιδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Πραγματικά η ιστορία αυτή δεν είχε καμία υπερβολή. Είναι ενδεικτική των δυσκολιών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα ανάπηρα παιδιά και οικογένειε του καθημερινά. Πώ λοιπόν αυτά τα παιδιά να δουν άσπρη μέρα και να προκόψουν. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά είναι η ελπίδα μα και θα πρέπει και από τη νέα κοινοβουλευτική θητεία ε, η η πρόεδρος Φοντερ Λάιεν ανέθεσε το χαρτοφυλάκιο σε έναν επίτροπο για μια συνολική σφαιρική στρατηγική για τα παιδιά. Ω εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παίξει κέριο ρόλο ώστε να εξασφαλίσει τήρηση των δικαιωμάτων όλων των παιδιών κατά την ανάπτυξη αυτή τη στρατηγική. Και η προγραμματισμένη εγγύηση για τα παιδιά επικεντρώνεται σε βασικέ υπηρεσίε δωρεάν παιδεία και υγεία αξιοπρεπού στέγασης και δωρεάν παιδικής μα. Αυτό είναι σημαντικό βήμα προ τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζουμε να εφαρμοστεί και από τα κράτη-μέλη. Εμείς, ε, η Eurochild, θα θέλαμε στο μέλλον να έχουμε και μια ευρωπαϊκή στρατηγική ε, του 2030 με συγκεκριμένο στόχο για τη μείωση της φτώχειας των παιδιών και θεωρούμε ότι τα παιδιά θα πρέπει να είναι ύψιστη προτεραιότητα του πολιτικού προγράμματος. Να θεσπιστεί αυτή η εγγύηση για τα παιδιά και να έχουμε μια αναβάθμιση των συστάσεων για των παιδιών και να έχουμε και συστάσεις του Συμβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα της επενδύσεις στα παιδιά. Ε, μόλις ολοκληρώσαμε την αξιολόγηση του 2019 για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Πρόκειται για μια έκθεση αξιολόγησης ε, 22 χώρων μελών. Η έκθεση της Eurochild επισημαίνει την έλλειψη προσοχής ε, του θέματος της παιδικής φτώχειας. Και μάλιστα ε, δεν έχουμε αρκετή συμμετοχή των παιδιών, οπότε και η παιδεία θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, περισσότερη στήριξη των οικογενειών και εναλλακτική ε, φροντίδα των κοινοτήτων. Θα πρέπει η ευημερία των παιδιών να περιληφθεί στην ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για, τις, για την ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών στις εκθέσεις αναχώρα Παρακαλώ ολοκληρώστε, λέει ο πρόεδρος. Και κλείνει το μικρόφωνο της κυρίας Πρέκα. Πάντως είμαστε ε, υπερήφανοι στη Eurochild που μέσω των συμβουλίων τα παιδιά μας ενημερώνουν για τις θέσεις τους και ελπίζουμε ότι και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα στο μέλλον θα έχουν ε, συμμετοχή των παιδιών με συγκροτημένο και διαρθρωμένο τόπο στη διαδικασία τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το βλέπετε το πρόβλημα του χρόνου. Πρέπει να τελειώσουμε στις 4.30 αυτό το πάνελ. Δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν όλοι όσοι το επιθυμούν. Διότι μακρηγορήσαμε και μας έφυγε ο χρόνος. Εδώ στο κοινοβούλιο μας είναι σημαντικό να το γνωρίζετε. Υπάρχει μια διακομματική ομάδα, έτσι λέγεται, ένα intergroup για τα δικαιώματα των παιδιών και των ανηλίκων. Και είναι δύο γυναίκες που είναι πάρα πολύ άξιες και γενναίες και πολύ στρατευμένες στην κατεύθυνση αυτή. Για να κάνει το κοινοβούλιο πολύ περισσότερα από το να μιλάει μόνο. Είναι η Χίλντε Βάουτμανς και η Κατερίνα Κινίτσι. Παρευρίσκονται και οι δύο και θα πάρουν πρώτες το λόγο. Ένα λεπτό όμως. Η κυρία Κινίτσι, πρώτα και μετά. Ένα λεπτάκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ λίγο πραγματικά γιατί πάρα πολλά θα θέλουμε να αλλά πρώτα, πρώτα να ευχαριστήσουμε όλους τους ομιλητέ και επίσης γυρίω τα παιδιά τα οποία μίλησαν και όσα παιδιά βρίσκονται στην αίθουσά μα. Όντως αυτή η στράτευση είναι για να εξασφαλίσουμε αυτή την συμμετοχή και αυτό έγινε και με το Intergroup για τα δικαιώματα των παιδιών και αυτό θέλουμε να το ανασυστήσουμε και είχαμε δουλέψει εκεί στην προηγούμενη ε, θητεία με τους άλλους ε, αντιπροέδρους και διάφορους βουλευτές συνάδελφους σήμερα. Είναι ιδιαίτερα σημαντική ημέρα, ε, εορτάζουμε και εορτάζουμε σημαίνει επίσης ότι θέλουμε να προσέξουμε τι γίνεται, να δούμε τι άλλο θα πρέπει να κάνουμε, να συσπηρωθούμε, γιατί είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία τα εκμεταλλεύονται, είναι στη φτώχεια, δουλεύουν, ε, ε τα εκμεταλλεύονται, είναι πάρα πολλά ε, βρέφη. Όλα αυτά είναι στην Ευρώπη και υφίστανται ακόμα πάρα πολύ βία. Οπότε, ε, κατακλείδη, να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε και κυρίως για αυτή την βία μέσω του Ιντερνετ. Η κυρία Βότμαν και μετά η κυρία Πρικμόν. Που συγγνώμη την ξέχασα, είναι και εκείνη στο Intergroup. Χωρίς μικρόφωνο κύριε Βότμαν. Α, τώρα δουλεύει. Καλησπέρα σας αγαπητά παιδιά και κυρία ε, Επίτροπε. Ε, η μισμενή μέρα είναι για τα παιδιά. Να σας πω μια ιστορία. Πριν από δύο χρόνια έχασα ε, ένα αγαπημένο πρόσωπο και ε, ε, ε, το γατάκι μου, τον Έλσονα, τον βρήκαν μέσα δύο ώρες γιατί χάλασα τον κόσμο στα social media και πήρα likes και πήρα και μηνύματα και τα λοιπά. Αλλά δεν βλέπω στο ίντερνετ να γίνεται χαμός για τις 10.000 ανηλίκους που έχουν χαθεί από τη μετανάστευση. 10.000, δεν τους ψάχνουμε, τα γατάκια τα ψάχνουμε. Πού είναι τα παιδιά, ουδής γνωρίζει και ουδής νοιάζεται. Αλλά θα πρέπει να ε, κάνουμε τέτοιες δράσεις, αναζητήσεις για τα παιδιά. Αυτή είναι η προτεραιότητα για τα 30 χρόνια της σύμβασης. Ε, να κάνουμε τον κόσμο μας ασφαλή κόσμο για όλα τα παιδιά μας και τα μεταναστόπουλα και τα προσφυγόπουλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρωτοβουλία, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η επέτειος. Είχα ετοιμάσει ομιλία, αλλά άκουσα τους νέους με τις συγκλονιστικές μαρτυρίες του και πραγματικά έθεσαν το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων. Ε, είδαμε τι προκλήσεις έχουμε ενώπιον μας, γιατί στην, ε, σε κάθε επέτειο ε, είναι ευκαιρία για γιορτή, κόβουμε και τούρτα, αλλά ουσιαστικά έχουν μείνει τα ψίχουλα στο σημερινό κόσμο για πολλού νέου. Οπότε θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση προς κυβερνήσει μα και πραγματικά θέλω να υπολογίσω σε εσά για να κρατήσετε αμύωτη την πίεση και την κινητοποίηση. Και ε, να στυλιτεύσουμε τι κυβερνήσει για την αδράνειά τους. Ένα παιδιά στα τέσσερα ζουν ε, στα κατόφλι ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Πολλές χώρες και η πατρίδα μου το Βέλγιο εξακολουθεί να ε, καρατά παιδιά στα πλαίσια της μεταναστευτικής πολιτικής ε, σε κέντρα, σε αντίθεση και καταστρατηγώντας την ε, Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Συνεχίστε λοιπόν την κινητοποίηση, γιατί πραγματικά οι πολιτικοί σας χρειάζονται, σας έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φέστη, ένα λεπτό. Ähm, Ευχαριστώ. Ε, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, σήμερα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια των δικαιωμάτων των παιδιών. Για ποιο λόγο όμως σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη και οι στατιστικές είναι πεντακάθαρες, ε, οι γάμοι με το στάνιο ε, αυξάνονται δραματικά όπως και ο κροτηριασμός των γεννητικών οργάνων 70.000 μόνο στη Γερμανία το 2018 και 800 καταναγκαστικοί γάμοι. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία. 70.000 και 800 γάμοι που δεν είναι τίποτα άλλο παρά ε, βιασμός ανηλίκων ε, που υποτίθεται ότι νομιμοποιείται. Αυτό στη Γερμανία και μόνο. Και αυτό θέλετε να το γιορτάζετε Ξέρουμε ότι στους καθολικούς δεν παντρεύονται τα παιδιά με το στανιό, ούτε στους Εβραίους, ούτε στους Βιδιστές, ούτε στους Προτεστάντες. Ε, ε, μόνο στο Ισλάμ γίνονται αυτά. Ε, αλλά πολλοί βουλευτές, κυρίως των Πρασίνων, των Αριστερών και των Σοσιαλιστών, κάνουν τα στραβά μάτια στη βία κατά των γυναικών και των παιδιών θεωρούν ότι αυτό έχει να κάνει με το φύλλο και ποτέ με τον πολιτισμό και την κουλτούρα. Αυτό που κάνουμε τα στραβά τα μάτια στο Τέλφορ, στο Oxfordshire και αλλού ε, κάνει τα παιδιά να υποφέρουν κάθε μέρα. Ξέρετε δεν έχετε χρόνο. Καθημερινά τα ζούμε αυτά και στην Κοπενχάγη και στο Βερολίνο και στο Αμβούργο. Αντί να γιορτάζετε να ντρέπεστε καλύτερα εδώ πέρα μέσα. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λέω και προς τους ενήλικες και προς τους νέους. Προσπαθήστε να ε, τηρείτε το χρόνο σας, αλλιώς αναφερείτε από άλλους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει και εμείς να το μαθαίνουμε και να δίνουμε το καλό παράδειγμα. Κύριε Φέστ, η κυρία Κέρα Μιράντα. Ευχαριστώ. Είμαι εδώ με τους συναδέλφους από ένα δίκτυο εκατοντάδων πανεπιστημίων και επιμορφώνουμε ε, τους επαγγελματίες για θέματα εκδημοκρατισμού και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ε, πρόσφατα είχαμε τη μελέτη για, στη Γενέβη για τα παιδιά και την παιδική φτώχεια. Θα σας ε, ενημερώσει ο συνάδελφος. Πάντως, παρόλο που έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κράτηση παιδιών μεταναστών σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετεί το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού, τουλάχιστον 330.000 παιδιά σε 8 χώρες βρίσκονται σε κέντρα κράτησης το κάθε χρόνο σε διάφορες χώρες. Οπότε θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό το γεγονός. Επίσης, ε, ζητήματα ψυχικής υγείας. Η στέρηση της ελευθερίας επιδεινώνει την υγεία και ειδικά την ψυχική υγεία και μπορεί να προκαλέσει νέα προβλήματα με το τραυματικό ε, στρες, άγχος, ε, κατάθλιψη και επίσης ε, η παράνομη αυτή κράτηση συνδέεται και με πρόωρο θάνατο παιδιών μετά την απελευθέρωσή τους. Θα πρέπει λοιπόν επίσης να φροντίσουμε πώς θα τους συμπαρασταθούμε για να αντιμετωπίσουν τα ψυχικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν μετά τα δράματα και τις τραγωδίες που έχουν ζήσει. Η κυρία Μπόνη. Ε, hello everybody. Ο κύριος Μπόνη μάλλον, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ε, και εγώ έχω κάνει το αυτό το μεταπτυχιακό των ανθρώπινων δικαιώματα και έχω εργαστεί στο μέτωπο των δικαιωμάτων LGBTI Κάποιος που λεγόταν ε, Μάθιου πήγε στους προσκόπους και ήταν στρατευμένος την ε, Έτζερ να κάνει κατά τον πλανήτη και όταν πήγε στο πρώτο του ε, στο πρώτο στρατόπεδο, στο πρώτο κάμπ των προσκόπων τους είπε ότι ήταν ομοφιλόφιλος και στην κατασκήνωση είχαν αρχίσει όμως τότε να τον χτυπούν μέχρι θανάτου έτσι νόμιζαν ότι ήταν και κλήθηκε η μητέρα του για να τον υποδεχτεί και θα έπρεπε να καταλήφθει η τασκήνωση αφού τον τιμώρησαν με αυτό το ξυλοκόπηση. Έπαθε κατάθλιψη και τελικά αυτοκτόνησε. Όμως δύο φορές πέθανε στην πραγματικότητα. 70% των ανθρώπων στην Πολωνία θέλουν να αυτοκτονήσουν. Ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι να κάνει τα δικαιώματα όλων των παιδιών. Bien. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Το 66, τα χάρ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί νέοι, είναι τιμή μου που παρίσταμε και έχω μια ερώτηση πρώτα πρώτα. Τώρα το 2019 έχουμε πάρα πολλούς νέους που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Παλαιστίνη, Συρία, Σομαλία, η Ουιγκούρ. Παρά το άρθρο 26 που λέει ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην παιδεία και τελειώνω την ερώτησή μου με αυτή την παρατήρηση. Αλλάζει ο κόσμος, αλλά η ανθρωπότητα πάει πίσω. Tom Belanger, puede ser 102. 102, Tom Belanger. Ονομάζομαι Τομ Belanger, είμαι 17 χρονών και πρέσβης στη δράση για τη Μεσόγειο. η ερώτηση είναι ταμπού. Τι κάνουμε με τα παιδιά που βρίσκονται σε καταβλήμους στη Συρία, στην Τουρκία και που κατηγορούνται ουσιαστικά για εγκλήματα που έχουν διαπράξει οι γονείς τους και έχουν αρκετά υποφέρει από την απομόνωση, από τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και παρόλα αυτά είναι καταδικασμένα να επιβιώσουν. Ας αλλάξουμε λοιπόν την κατάσταση, να μην πληρώνουν τα σπασμένα και τα λάθη των γονιών τους. Σας άκουσα κυρία Γιώροβα με πολύ προσοχή. Αλλά για να έχει νόημα η ομιλία σας και για να έχει νόημα αυτή η επέτειος θα πρέπει να επαναπατρίσουμε τα παιδιά αυτά και να σεβαστούμε τα δικαιώματά τους. Η Ευρώπη έχει, έχει καθήκον να προστατεύσει τα παιδιά αυτά και τα δικαιώματά τους για να αποκτήσουν εμπιστοσύνη και να επανασυμφιλειωθούν με τις ε, αξίε της δημοκρατίας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η σιωπή σα πραγματικά είναι επέσχυντη. Και όπως είπε και η Άχρατ, ας, ας αφήσουμε τα παιδιά να είναι παιδιά. Να μην τα, αφήνουμε ως, ε, να μην τα αντιμετωπίζουμε ως ορολογιακές βόμβες. Είναι παιδιά όπως και εμείς. Ας δράσουμε επιτέλους. Σας παρακαλώ. Bien sûr, merci. Michel Mates. Mates. Michel Mates. Στο 242. Εγώ είμαι, ναι. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Μάικελ από την Συμμαχία για την Παιδική Ηλικία. Την πρώτη μέρα ε, ανάληψη των καθηκόντων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, διοργανώσαμε μια συναυλία παιδιών που έπαιξαν και τραγούδησαν ε, τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το 2020 θα κάνουμε το ίδιο την 1η Σεπτεμβρίου. Ας καθιερώσουμε αυτή την τελετή, να αρχίζει τις εργασίες του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με αυτόν τον τρόπο με τα παιδιά. Εγώ είμαι από τις κάτω χώρες και την πρώτη ημέρα έναρξης των κοινοβουλευτικών εργασιών όταν ανοίγει η Βουλή το γιορτάζουμε. Ας το γιορτάζουμε και εδώ για τους πολίτες και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 1η Σεπτεμβρίου να επαναλάβουμε ε, αυτή τη δράση και να παίξουν τα παιδιά τον ύμνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Thank Ευχαριστώ πολύ. Άννα You Thank you so much. Uh, ευχαριστώ πολύ. Έχω ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις, αλλά δεν θα τις διαβάσω. Θέλω ένα σχόλιο για όλους σας. Ξέρετε, γι' αυτό πολιτεύομαι, για να δώσω φωνή στους νέους στο μέλλον και σας ευχαριστώ που φέρετε την ενέργειά σας εδώ στην Ολομέλεια αλλά και με πραγματικές ερετήσεις και περιεχόμενο και θέλω να σας ζητήσω να διατηρήσετε όλο αυτό το σφρίγος και το σθένος γιατί όλα αυτά τονίζουν πραγματικά ότι ε, ε, ε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε την διακήρυξη της Βουδα... του, του Βουκουρεστίου. Γιατί δεν θα πρέπει μόνο οι νέοι να ασχολούνται με την πολιτική, οι νέοι ενήλικοι, αλλά και τα παιδιά. Εγώ ακούω καθημερινά ότι είμαι πολύ νέα για να ανακατεύομαι στην πολιτική. Μια ερώτηση έχω μόνο για τα κορίτσια του πάνελ μπορείτε να μας πείτε σας παρακαλώ πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο τα θέματα των παιδιών να συντονίσουμε τη φωνή μας, να τη φέρουμε πιο κοντά σε εσένα για να ακούγεται και η δική σας φωνή. Ευχαριστώ. Ιβάνα Νόα, 70. Ιβάνα Νόα, στο 70. Ιβάνα Νόα, 16 ετών. Πιστεύω ότι κάθε παιδί θα πρέπει να έχει μια ευκαιρία η γενιά μας κινείται γρήγορα και μαθαίνει πολύ γρήγορα. Θα πρέπει λοιπόν να, ενισχύσετε τα παιδιά δίνοντας την ευκαιρία να μιλήσουν, να τους εξασφαλίσετε ασφαλές μέρος ώστε να μπορούν ελεύθερα να πούν την γνώμη τους. Η Σάλλη Γκορνίτσκα, η αναπληρωτήρια γενική διευθύντρια της UNICEF, είπε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι το καθιστικό των νέων. Εκεί που περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να μπορούν τα παιδιά να εκφράσουν τη γνώμη τους. Θέλουν μια πλατφόρμα για να μπορούν να πούν τι νιώθουν, να νιώθουν ασφάλεια. Θα πρέπει να δώσουμε μέλλον στα παιδιά, γιατί όταν δίνουμε μέλλον στα παιδιά θα πάρουν αυτή την ευκαιρία. Είμαι ε, σκηνοθέτης και πιστεύω ότι με μια κάμερα μπορεί να ενεργοποιηθεί το δυναμικό των παιδιών. Και με ένα πινέλο μπορούμε να δημιουργήσουμε τον επόμενο Παύλο Πικάσο. Ευχαριστώ. Thank you Ο Μάθιου Πάτεν. Ευχαριστώ. Μάθιο Πάτεν. Είμαι 57, αλλά νιώσω θα σαν 18. Ακούσαμε πολλά θερμά από εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού αλλά δεν θα πρέπει να ξεγελαστείτε από την κολακία και το δωρεάν καφέ. Τα τελευταία χρόνια πολλές υποσχέσεις έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα παιδιά, αλλά δεν τη στήρισε. Και ο κύκλος της παιδικής φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αλλάξει παρά ελάχιστα. Οπότε μερικά πράγματα μόνο μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον. Καταρχήν, σηκώστε τα χέρια. Ποιο από εσά έχει συναντήσει την Εύα Κόπατ που είναι η Ευρωπαία αρμόδια για το θέμα αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σηκώστε το χέρι δεν τη γνώρισε. Θα πρέπει να βγει από το γραφείο της, να έρθει σε επαφή μαζί σας, να δείτε τι συμβαίνει επί τόπου, να απαιτήσετε να έρθει να σας συναντήσει. Αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεδομένου ότι τα παιδιά και οι οικογένειες από εθνικέ και άλλες μειονότητες ε, πλήττονται κυρίως από τη φτώχεια, θα πρέπει να τους δώσουμε ένα ρόλο σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι θεσμικά ρατσιστικό. Σε όποιους και, αν, οποιους ε, και αν μίλησε μέχρι στιγμής ήταν λευκός. Θα πρέπει λοιπόν και οι μειονότητες ε, να αποκτήσουν θέση εξουσίας για να μπορούν να μιλήσουν, να εργαστούν, να διαβιώσουν και να ηγηθούν. Ευχαριστώ. Εις αλτίντας. αλτίντας. 154 ή 155. Φωτογράφος και δάσκαλος. Έχετε το λόγο. Γεια σας, ονομάζομαι Ίσα. Προέρχομαι από την ε, Γερμανία με τουρκική καταγωγή. Είμαι καθηγήτρια ή δασκάλα και θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την κατάσταση των παιδιών που έχουν θυγεί από πολιτικά ζητήματα που εκκρεμούν στην Τουρκία πολύ καιρό. Στατιστικά έχουμε 11.000 γυναίκες και 780 παιδιά που είναι φυλακισμένοι σήμερα στην Τουρκία. Ήρθαμε εδώ να γιορτάσουμε την επέτειο των δικαιωμάτων παιδιών που προσυπέρεψε η Τουρκία πριν από 30 χρόνια, αλλά από φέτος 2019 παιδιά κάτω των 6 βρίσκονται στην φυλακή με τις μητέρα τους και χιλιάδες παιδιών δεν απολάβουν των θεμελιωδών δικαιωμάτων οι γονεί του, Είναι στην αντιπολίτευση και γι' αυτό και φυλακίζονται. Σας ερωτώ. Έχει αναλυθεί η κατάσταση. Για yeah. αυτά τα πρόσωπα προσπάθησε κανείς να τους βοηθήσει. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι λύση μπορεί να υπάρξει. Ευχαριστώ. Η Ανίτα Νιάμε. Ε, καλησπέρα σε όλους. Ανίτα, από την Κάνα κατάγομαι. Ε, είμαι μέλος του Φλαμαδικού Συμβουλίου Νεολαίας για το Βέλιο Χαίρομαι που οι πολιτικοί και σημαντικοί άνθρωποι έρχονται να μας μιλήσουν. Αλλά ρωτιέμαι όμως τι γίνεται με τις συμβουλές που δίνουμε εμείς σε όσους παίρνουν τις αποφάσεις. Όλοι λέτε ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε ε, και να μιλάμε δυνατά, χωρίς φόβο. Μιλάμε δυνατά, χωρίς φόβο και συμμετέχουμε. Αλλά εσείς αυτά που σας αναλογούν τα κάνετε. Γιατί εσείς μας διδάσκετε να σηκωθούμε, να υψώσουμε τη φωνή μας και να συμμετέχουμε. Όλα αυτά που μας ε, λέτε τα κάνετε εσείς. Πώς βεβαιώνεστε ότι αυτά που σας προτείνουν τα παιδιά ε, βρίσκουν το δρόμο τους στις δικές σας εργασίες. Ποιες είναι οι δράσεις που αναλαμβάνετε για να σπάσουν αυτά τα εμπόδια. Ευχαριστώ. Freya Freeman Taylor. Freya Freeman Taylor. Στη θέση 354. Έδρανα 354. Μάθιου Μπριένσενς Στο έδρανο 334, 335. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτή την καταπληκτική σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και να επιθυμίσω το άρθρο 3 που προβλέπει ότι σε όλες τις ε, αποφάσεις ε, που αφορούν τα παιδιά ε, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού. Παρ' όλα αυτά με προβληματίζει, με ανησυχεί αυτό που άκουσα και στην έναρξη της διάσκεψης αλλά και ε, από την ομιλία της UNICEF. Τίποτα δεν αναφέρθηκε ούτε μία κουβέντα για το άρθρο 7 το άρθρο που αφορά τη γέννηση του παιδιού. Και από τη στιγμή που, όπως λέει η UNICEF, ε, το, δικαίωμα, ε, το παιδί έχει δικαίωμα σε όνομα, σε ηθαγένεια και σε ταυτότητα, θα πρέπει να, να πει ότι το παιδί στο μέτρο του δυνατού θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τους βιολογικούς τους γονείς και να ανατραφεί από αυτούς. Και όταν μιλούμε για τους γονείς, ενώ τους βιολογικούς φυσικά γονείς, γνωρίζουμε όμως όλοι σήμερα ότι πολύ συχνά οικειοθελώς τα παιδιά χωρίζονται από τους γονείς τους και τους δύο ή μόνο τον πατέρα τους ή τη μητέρα τους. Επίσης έχουμε και την βαρέθετη μητρότητα το 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε αυτή την πρακτική. Παρ' όλα αυτά συνεχίζεται. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να τηρηθεί αυτό, αυτή η Ευρωπαϊκή Νομοθετική Διάταξη που συνάδηκε με το άρθρο 7 της Διεθνούς Σύμβασης για, το, για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σας ευχαριστώ θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουν πολύ περισσότεροι, αλλά βλέπετε πόσο περίπλοκο είναι να προεδρεύεις. Πάρα πολύ. Παρευρίσκεται η πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, η ε, ε, Λούση ε, Λετσινγκα. Είναι πολύ καλό και πολύ σημαντικό να την ακούσουμε. Και μετά θα απαντήσει το πάνελ. Bien. Primero las respuestas del panel y luego Lucy, Lucy Μάλλον πρώτα ε, τα μέλη του πάνελ και μετά η Λούση Μετσίνγκια. Πολύ σύντομα όμως τις απαντήσεις παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τους διοργανωτές αυτής της διάσκεψης ψηλοεπέδου επευκαιρία της 30ης επαιτίου της ε, σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Ήταν η πρώτη διεθνή ε, σύμβαση που αναγνώρισε τα παιδιά ως πραγματικούς δικαιούχους και φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτή η σύμβαση συνέβαλε σε ρηξικέλευτες αλλαγέ ε, στο πώ βλέπουμε τα παιδιά στι κοινωνίε μας. Βέβαια, 30 χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ εξακολουθούν ε, να παραμένουν πολλέ προκλήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τα νεαρά μέλη του πάνελ που μα παρουσίασαν τι ιστορίε του, την ε, Ακράτ, τη Ράινα και τον Σίντι και όλους άλλου νεαρούς. Οι φωνές τους είναι πολύ σημαντικέ και του ευχαριστώ θερμά για τι παρεμβάσει του. Η συμμετοχή των νέων στη διαδικασία λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα των ευάλων των νέων, όπω είναι των νέων που είναι παιδιά μεταναστών ε, Ρωμά, που έχουν εμπλακεί σε σειράξει ή έχουν αναπηρίε, είναι το σημαντικότερο χέγγιο για την προστασία των, ε, των δικαιωμάτων των παιδιών και η προστασία του από, από την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό. Η σύμβαση προβλέπει το δικαίωμα των παιδιών και των νεαρών να εκφράζουν ελεύθερα τι απόψει του για θέματα που του αφορούν και να λαμβάνονται επίση δεόντω υπόψη αυτέ οι απόψει. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα δικαιώματα να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αφουγκραζόμαστε ε, τα παιδιά. Ακούσαμε τη Ράινα που είναι μέλος ομάδας της Γκρέτα Θούμπερκ και να έκκληση να δράσουμε τώρα για να προστατεύσουμε το δικαίωμα σε ένα καθαρό περιβάλλον. Και μάλιστα το κίνημα της Γκρέτας ε, ε, έχει κινητοποιήσει εκατομμύρια παιδιά που θέλουν να εισακουστεί η φωνή του ε, και τα αιτήματά του και τα δικά μου παιδιά συμμετέχουν σε αυτές τις απεργίες για το περιβάλλον. Οι προκλήσει τη κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει σημαντικά τα παιδιά σε όλο τον κόσμο και θα πρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσει. Το 2019 θα είναι η χρονιά που η πρόοδος, ε, θα αξιολογηθεί η πρόοδος για την ε, υλοποίηση των στόχων του 2030 που ζητά ένα κόσμο που θα επενδύει στα παιδιά και που κάθε παιδί θα ζει χωρίς ε, βία και χωρίς εκμετάλλευση. Επίσης έχουμε τον ψηφιακό κόσμο και τις τεχνολογίες πληροφορίας και τεχνολογίες που επηρεάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών. Ο ψηφιακός κόσμος προσφέρει, προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες και γνώση, αλλά θα πρέπει να είναι προσιτό σε όλα τα παιδιά, χωρί καμία διάκριση. Ταυτόχρονα έχουμε και μίσο που το ίντερνετ και ο ψηφιακό κόσμο είναι πολύ επικίνδυνο για τα παιδιά, με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την παιδική πορνογραφία. Είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά και να εξασφαλίσουμε αξιόπιστε και σωστέ ακριβεί πληροφορίε για τα θέματα που αναζητούν. Επίση, λίγα λόγια για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, στην οποία προεδρεύω. Ασχοληθήκαμε με θέματα διασυνοριακού οικογενειακού δικαίου και την αναδιατύπωση ε, του κανονισμού Βρυξέλλες 2 για την ε, γονική μέρημνα. Λαβάζουμε υπόψη το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού και τη σχέση με τους γονείς εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα που χρειάζονται τα παιδιά. Επίσης, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα πρέπει να φροντίσει ώστε και τα θετά παιδιά να έχουν άμεση πρόσβαση σε δικαστική διαδικασία που να εξασφαλίζει επίσης μια ασφαλή και σταθερή κατάσταση. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας και την προσοχή σας. Επαναλαμβάνω ότι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα κοφεύσουμε στα αιτήματά σας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιταχύνουμε τις προσπάθειες και, στα για τα δικαιώματα των παιδιών και την προστασία τους και για την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει φυσικά να ε, ακούσουμε πρώτα τη φωνή των παιδιών και μετά να κάνουμε και εμείς το καθήκον μας ως πολιτικοί και να περάσουμε στη δράση. Ευχαριστώ. θέλαμε τώρα να μπορούν να απαντήσουν και τα μέλη του πάνελ. Θα σας στείλουμε γραπτός ε, τις απαντήσεις γιατί δεν προλαβαίνουμε. Θα δούμε ένα βίντεο τώρα της UNICEF που δείχνει πώς συνεργάζονται ε, με προγράμματα, Ευρωπαϊκή Ένωση με τη UNICEF. Ακριβώς σε ένα ε, πρόγραμμα για να δούμε ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα και οι προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Θα δείτε πώς λειτουργήσε αυτό. Πριν δούμε αυτό το βίντεο, θα ήθελα να πω ότι σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας που δεν το βάζετε κάτω που δεν παραδίδεστε, που απαιτείτε και σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που θα κάνετε πάρα πολύ σύντομα. Να δούμε λοιπόν το βίντεο. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Αρχίζει λίγο το δεύτερο πάνελ. on va... Alors, on... Λοιπόν, est-ce que je peux... Μήπως θα μπορούσα να σας ζητήσω... Ξέρω ότι ήσασταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Καθίστε πάλι. C'est un peu plus soft que le marteau. ouais, non, mais c'est plus soft que le marteau. Λοιπόν, καθίστε σας παρακαλώ. Και όσοι θέλετε να αποχωρήσετε, αποχωρήστε ησύχως. Έξω ιδιωτικές συνομιλίες παρακαλώ. Για να δώσουμε την ευκαιρία σε όσους παραμείνουν και όσες να ακούσουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξέρω ότι χρειάστηκε να συγκεντρωθείτε πολύ για το πρώτο πάνελ, αλλά θα περάσουμε στο δεύτερο πάνελ που θα ασχοληθεί με το όνειρο. Ακούγοντας το πρώτο πάνελ πραγματικά ονειρευόμουν εδώ στην αίθουσα να έχουμε κατά τη διάρκεια των συνόδων της Ολομέλειας το ίδιο πνεύμα. Έτσι ένα ανοιχτό πνεύμα, ένα πνεύμα αλληλεγγύης, ανεκτικότητας οραματικό που καμιά φορά νομίζω λείπει από τους νέους, από τους, μάλλον τους ε, ε, ενηλίκους εκλεγμένους εδώ βουλευτές. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε εδώ εκπροσώπους και αν ήσασταν εσείς παρόντες θα είχαμε κερδίσει ένα κείμενο το οποίο κείμενο είχε να κάνει με τη διάσωση στη θάλασσα, διάσωση των μεταναστών. Δυστυχώς όμως επειδή δεν είχαμε το δικό σας πνεύμα εδώ να πριτανεύει, επειδή κάποιοι από το κοινοβούλιο εδώ δεν είχαν αυτό το όραμα για ένα καλύτερο κόσμο, χάσαμε αυτή την ψηφοφορία για το κείμενο αυτό με δύο ψήφους διαφορά. Και πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε όλοι. Θα σας παρουσιάσω τα μέλη του πάνελ πάρα πολύ γρήγορα. Ε, ακούσαμε προηγουμένως ότι γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της σύμβασης αυτής. Μπορεί να δει κανεί λοιπόν το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Εγώ είμαι φύση αισιόδοξη και θέλω να το βλέπω μισογεμάτο. Αλλά κυρίως θέλω να το γεμίσω και το υπόλοιπο και εδώ μιλώ για τις προκλήσεις που δεν αντιμετωπίζουμε. Εγκλισμός των παιδιών. Πάνω από 1,5 εκατομμύρια κρατούνται σε φυλακές παιδιά σήμερα. Μιλήσαμε για τη μετανάστευση. Τα παιδιά που είναι τα θύματα αυτής της μετανάστευσης. Που στη χειρότερη περίπτωση πνίγονται στη Μεσόγειο ή χάνουν αλλού τη ζωή τους στο δρόμο. Ή ε, είναι γεμάτο παγίδες ε, ε, αυτό το μονοπάτι που παίρνουν και ο δρόμος τους τους κάνει να ζουν φρικαλαιότητες και φτάνουν στην Ευρώπη για να κλειστούν σε κάποια κλειστά κέντρα. Μιλήσαμε επίσης για την παιδική εργασία, μιλήσαμε και για τις μελλοντικέ προκλήσεις αλλά και για τις σημερινές, για την προστασία των παιδιών, για την προστασία από την κλιματική αλλαγή. Συχνά μιλούμε για την υπερθέρμανση του πλανήτη αλλά όχι θέματα περιβαλλοντικά, για την προστασία των παιδιών από ουσίες που ε, ε, προκαλούν διαταραχές στο ενδοκρινικό σύστημα. Σήμερα τα παιδιά μας έρχονται αντιμέτωπα με προϊόντα και ουσίες που δεν ξέρουν ότι θα βλάψουν την υγεία τους. Ε, είναι αυτά θέματα επίσης σημαντικά όπως και η ψηφιακή τεχνολογία που μπορεί να είναι θετική και είδαμε στην καμπάνια τι έγινε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε ε, θετικά την ψηφιακή τεχνολογία για να κάνουμε και πάρα πολλά καλά αλλά μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει για εκφοβισμό, για bullying, για παρενόχληση ή για να σπέρνει ζυζάνια και να βάζει κακές ιδέες στα μυαλά των παιδιών ενηλίκων. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν εδώ στο Κοινοβούλιο τα αντιμετωπίζουμε, αγωνιζόμαστε δεν αγωνιζόμαστε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Ε, ε, πάντως χρειάζεται συνοχή σε αυτό τον αγώνα, γιατί καμιά φορά λειτουργούμε παράλληλα, κάθετα, σε δομές απομονωμένες. Μιλάμε ε, για τα δικαιώματα των παιδιών, αλλά όχι για τις πολιτικές που άμεσα ή έμεσα έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα. Χθες ήμουν στην Αφρική και εκεί μιλήσαμε για ένα θέμα για το οποίο δεν μιλάει κανείς εδώ, που είναι οι ευρωπαϊκές εξαγωγές από βουτυρωμένου γάλακτος στην Αφρική και μάλιστα στη Δυτική Αφρική. Και θα μου πείτε, μα τώρα τι μας ε, τσαμπουνάς. Ε, υπάρχουν γαλλικές εταιρείες, ευρωπαϊκές εταιρείες, δανώνες, Nestlé, που βγάζουν τρελά λεφτά στην Ευρώπη και πηγαίνουν στην Αφρική και πάνε να πουλήσουν γάλα, αλλά δεν είναι γάλα, είναι γάλα από όπου έχουν βγάλει το βούτυρο για να μπορέσουν να το ακριβο... πουλήσουν ακριβά στην Κίνα και μετά βάζουν φινικέλαιο στο γάλα αυτό και το πουλούν στην Αφρική σε πληθυσμούς φτωχούς που πληρώνουν αυτό το γάλα 40% φθηνότερο. κάνοντας αυτό καταστρέφουν τους εντόπιους παραγωγούς που βγάζουν καλό γάλα και στην Κάνα και αλλού γεμίζουν τις τσέπες των πολυεθνικών και τα, κυρίως έρχονται ε, να πλήξουν ε, την υγεία των παιδιών στην Αφρική γιατί δεν τρέφονται με καλά προϊόντα. Ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτό θα πρέπει να στραφούμε. Να έχουμε συνεκτικές και συνεπείς πολιτικές, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των παιδιών, όχι γενικά και αόριστα, αλλά σε όλες τις πολιτικές που μπορούν και έμεσα να επιτεθούν σε αυτό το θεμελιώδη δικαίωμα που είναι δικαίωμα στην υγιεινή τροφή και δικαίωμα στο να έχεις γονεί που να δουλεύουν και να μπορούν να σου δώσουν υγεία και παιδεία. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν μια παγκόσμια συνολική προσέγγιση και στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα συζητούμε αυτά και ευχαριστούμε τους βουλευτές που είναι μέλη εκεί. Ανθρώπινα δικαιώματα, ε, γυναικεία δικαιώματα, δικαιώματα του παιδιού, όλα αυτά μας απασχολούν ευρύτερα. Για να συζητήσουμε λοιπόν για αυτά τα όνειρα, γιατί για όνειρα πρόκειται και για οράματα και πραγματικά μεγαλώνοντας θα ήθελα πάρα πολύ να διατηρήσουμε αυτά τα παιδικά μας όνειρα και να αγωνιζόμαστε για αυτά. Ε, έχω τη χαρά λοιπόν σε αυτό το δεύτερο πάνελ να έχω εδώ την κυρία Σίρλεϊ Αγιοκόρ Μποτσουέι που είναι υπουργό Εξωτερικών της Γκάνας. Επίσης έχω τη χαρά να υποδέχομαι τη Μαρία που έχει το ίδιο όνομα με μένα ε, από την Ουγγάντα. είναι 14 ετών. Επίσης την κυρία Σαρλότ Πετρί Γκορνίτσκα, που είναι αναπληρώτρια εκτελεστική διευθύντρια της UNICEF. Επίσης καλωσορίζω τον Μπερεκέτ, 16 ετών, από την Αιθιοπία που ζει όμως στην Γκάνα, αν δεν απατώμε, και τέλος τη Βελίνα Τοντόροβα που είναι Αντιπρόεδρος Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ. Θέλω να δώσω αμέσως το λόγο στη συνάδελφο Υπουργό Εξωτερικών της Γκάνα. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Πολύ Μαρία. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και ιδίω τα παιδιά, τους ηγέτες του μέλλοντος. Χαιρετισμούς από τα παιδιά της Γκάνας. Μαζί σας, σε εμάς ποντάρουν, ούτω ώστε να γίνει ο κόσμος καλύτερος μια μέρα. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση, για την ευκαιρία που μας προσφέρετε να συμμετάσχουμε ε, στην, ε, στο σημερινό εορτασμό της Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού. Και επίση ε, να ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί οργάνωσε αυτή την εκδήλωση ορόσημου και έτσι αποδεικνύει την στράτευσή του για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Πριν από τρεις δεκαετίες η Γκάνα υποσχέθηκε και δεσμεύθηκε να προστατεύει τα δικαιώματα των ε, παιδιών και κύρωσε την σύμβαση του ΟΗΕ, την σχετική. Και έτσι κατηγορούνται κάποια δικαιώματα των παιδιών γιατί πρόκειται για ευάλωτα πρόσωπα. Αυτά τα δικαιώματα καλύπτουν το δικαίωμα στο όνειρο, στην ε, ανάπτυξη, στο παιχνίδι, στην αξιοπρέπεια, στην μάθηση. Και σχεδόν 30 χρόνια από τότε που τέθηκε σε και συνθήκη τη Δευτέρα Σεπτεμβρίου του 1990 αναγνωρίζεται όπως η ευρύτερα κυρωμένη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ιστορία. Έτσι εμπνεύτηκαν οι κυβερνήσεις να αλλάξουν την νομοθεσία, να δώσουν πόρους στην ε, παιδεία για τα παιδιά, στην ε, υγειονομική κάλυψη, σε προστασία από εκμετάλλευση και βία. Επίσης, έτσι βρέθηκε μια πλατφόρμα για να ακούγεται η φωνή του παιδιού στην κοινωνία. Παρά αυτά τα βήματα πρώτα για την προστασία και πρόθεση του παιδιών η σύμβαση δεν έχει πλήρως εφαρμοστεί ούτε έχει ενταχθεί σε κρατικές πολιτικές και προγράμματα επίσης. Οι διατάξεις τη συνθήκη δεν είναι ευρέως γνωστέ, ούτε κατανοητέ. Εκατομμύρια παιδιών σε όλο τον κόσμο υφίστανται βία παραβίαση των δικαιωμάτων τους με γάμους αναγκαστικούς με εξαναγκαστική εργασία και επικίνδυνη εργασία δεν υπάρχει και κάλυψη μπαίνουν τα παιδιά στα ίδια κελιά φυλακής με ενήλικες όλα τα παγκόσμια προβλήματα ε, όπως η αργή του κλίματος, η πόλεμη, η τρομοκρατία, η ανασφάλεια και όλες τις σκοτεινές πτυχές ε, του ψηφιακού κόσμου έχουν επιδεινώσει τα προβλήματα των παιδιών. Όλα αυτά όμως δεν θα πρέπει να μας φέρνουν απελπισία. Θα πρέπει να είναι κίνητρο, μας φέρνουν αποφασιστικότητα για να συνεχίζεται το όραμά μας και η στράτευσή μας ότι θα υλοποιηθούν όσα οι ηγέτες το 1989 είχαν στο μυαλό όταν έφτιαξαν την ε, σύμβαση. Θα πρέπει πλήρως η σύμβαση να αποτελέσει τμήμα του εθνικού θεματολογίου. Θα πρέπει να έχει κάθε παιδί το δικαίωμα στο όνειρο να μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους άσχετα από φίλο, φιλή ή θρησκεία. Θα πρέπει κάθε ευκαιρία να την εκμεταλλευτούμε ούτω ώστε να μειωθούν οι απειλέ βάρο των παιδιών και θα πρέπει η πρόδοση τεχνολογίας να αξιοποιηθεί υπέρ του παιδιού και οι βασικοί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αυτή θα πρέπει να αναλάβουν δράση για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα παραβιάζονται τα δικαιώματα των παιδιών κυβερνήσεις, ε, αυτοί που διαμορφώνουν τους ε, πολιτικές, γονείς, ε, όσοι επιμελούνται ε, τα παιδιά όλοι όλοι οι ενήλικοι ενωμένοι να εξασφαλίσουν ότι οι στόχοι των βιώσιμων στόχων ανάπτυξης πρόκειται να βοηθήσουν και ήμουνα και εγώ νεαρή μητέρα στο παρελθόν και ήθελα τα παιδιά μου να τα μεταχειρίζουμε σαν ε, πρόσωπα με συγκεκριμένες συνθήκες και το ότι θα έπρεπε να έχουν τη σωστή ανατροφή και επίσης θα έπρεπε το περιβάλλον να ήταν φιλικό στο παιδί και να ακούγεται η φωνή του παιδιού. Ε, είχαν φωνή τώρα, σίγουρα θέλουν ε, τα παιδιά να συμμετέχουν στις συζητήσεις. Θέλουν να ακούγεται η γνώμη τους. πολύ σε όλο τον ε, κόσμο υποτιμούν αυτό το στοιχείο της σχέσης παιδιού γονέα. Όμως οι ενήλικοι και οι γονείς επηρεάζουν ε, τα παιδιά γιατί ε, αφορά αυτή η επιρροή θέματα τη ζωή των παιδιών. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ συναρπαστική η συζήτηση με το θέμα μα του ότι κάθε παιδί έχει το δικό το όνειρο. Και έχουμε και δύο παιδιά εδώ που θα μιλήσουν σχετικά με το θέμα, σχετικά με την άμεση επίδραση στην καλοπταχείριση των παιδιών για εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο. Ευελπιστώ ότι τα συμπεράσματά μας θα είναι ενθάρρυνση προς κυβερνήσεις και προς τους ε, βασικούς παράγοντες που εμπλέκονται ούτω ώστε να θωρακιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών παντού στον κόσμο και συμπερασματικά θέλω να σα πω ότι μια που είμαστε η πρώτη χώρα που κύρωσε τη συνθήκη η Γκάνα έχει δεσμευτεί υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών και αυτό συνεχίζεται με την αποφασιστικότητά μα να έχουμε ε, ένα καλά δομημένο ε, σύστημα κοινωνική πρόνοια ε, τα παιδιά και να τα προστατεύουμε από κακομεταχείριση ε, και από κάθε κακό. Επίσης έχουμε κατάλληλη νομοθεσία ε, ούτως ώστε να μην υφίστανται τα παιδιά στη χώρα μας σωματικές ε, τιμωρίες, βία στην οικογένεια και σεξουαλική εκμετάλλευση και παρανομή εργασία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Θα δώσω αμέσως το λόγο στη Μαρία. Έχεις το λόγο Μαρία. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Ονομάζομαι Ναζίουα Μαρία Γκορέτ από την επαρχία Μπουίκβε της Ουγγάντα. Είμαι νεαρή γιατί είμαι μέλος του Παιδικού Κοινοβουλίου και είμαι καταθουσιασμένη που γιορτάζουμε μαζί την 30η επέτειο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε αυτή τη διάσκεψη υψηλού επίπεδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως είπα, είμαι νεαρή ηγέτης και ο ρόλος μου ως ε, βουλευτής του Παιδικού Κοινοβουλίου είναι να δώσω φωνή σε παιδιά που δεν μπορούν να μιλήσουν για τα προβλήματα που τα ταλανίζουν. Ε, τα παιδιά στην Ουγγάντα πολλές φορές ντρέπονται να μιλήσουν με τους ενήλικες για τα προβλήματά τους. Παρόλο που είναι εύκολο να μοιραστούν μαζί μας με τους νεαρούς ηγέτες ε, αυτά που, τα, που τους ταλαιπωρούν. Και έτσι όταν ένα ε, παιδί μας λέει ένα πρόβλημα, εμείς το συζητούμε στο παιδικό κοινοβούλιο, έχουμε συζητήσεις και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις για τα προβλήματα. Ε, μετά διαβιβάζουμε τα προβλήματα και τις λύσεις στην Επιτροπή ενηλίκων και περιμένουμε να αναλάβουν κάποιες δράσεις. Και μάλιστα δίνουμε σε αυτή την Επιτροπή των Ενηλίκων ένα χρόνο, κάποιο χρόνο για να δράσει και αν διαπιστώσουμε ότι αυτή η Επιτροπή των Ενηλίκων χρόνο τριβεί, προσπαθούμε να ρωτήσουμε και να μάθουμε τους λόγους αυτής της αδράνειας και της καθυστέρησης και διαπιστώνουμε ότι παρόλο που έχουν γίνει πολλά πράγματα εξακολουθούμε να έχουμε φαινόμενα βίας κατά των παιδιών. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα λοιπόν για να σταματήσει η βία εις βάρος των παιδιών. Οι λόγοι που δίνω τη μάχη για να σταματήσει η βία κατά των παιδιών είναι εξή. Καταρχήν, τα παιδιά είναι η μελλοντική γενιά και αν παραβιαστούν τα δικαιώματά τους δεν θα έχουμε ένα καλό μέλλον. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί στερηθεί το δικαίωμα στην παιδεία, αυτό το παιδί δεν θα γίνει ποτέ κάποιος, δεν θα προκόψει. Οπότε φανταστείτε μία γενιά με παιδιά που δεν θα έχουν μορφωθεί, που δεν ε, θα έχουν καταρτιστεί. Θα πρέπει λοιπόν τα παιδιά να απολαύσουν τα δικαιώματά τους, να μπορέσουν να τα ασκήσουν για να έχουμε σωστό μέλλον. Επίσης, έχω αδέρφια, αδερφούς και μία αδερφή. Αν δεν δώσω λοιπόν μάχη για αυτούς, ε, για να καταργηθεί η βία, η σεξουαλική και η θυσία των παιδιών, κάποια στιγμή μπορεί και εμείς να γίνουμε θύματα, εγώ και τα αδέρφια μου, θύματα αυτής της σεξουαλικής βίας. Οπότε, για να αποτρέψουμε τέτοια φαινόμενα, θα πρέπει να συνεχίσουμε τη μάχη. Κάτι άλλο που συμβαίνει είναι αν τα δικαιώματα ενός παιδιού παραβιαστούν ε, και παρόλα αυτά μείνει αβοήθητο, το παιδί αυτό θα μεγαλώσει και θα νομίζει ότι είναι ok και δεν υπάρχει πρόβλημα να παραβιάσει τα δικαιώματα των άλλων. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε λοιπόν ένα παιδί να πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το να παραβιάζονται τα δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τον αγώνα μας για να τεθεί ένα τέρμα στη βία κατά των παιδιών. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά που είναι θύματα βίας για να μην μείνουμε την εντύπωση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να παραπιάζονται τα δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τη μάχη. Επίσης θα ήθελα να καλέσω όλους οι ενδιαφερόμενους και τα παιδιά, τους πολιτικούς ηγέτες, τους δασκάλους, θρησκευτικούς ε, οι αρχηγούς να ενώσουν τα χέρια τους, να συνεργαστούν για να δώσουμε ένα τέρμα στη βία γιατί χρειάζεται ο ενωμένο ο κόσμος για να δώσουμε ένα τέρμα στη βία και ο αγώνας θα ξεκινήσει από εσά, από εμένα και ε, εσάς. Γι' αυτό θα ήθελα να σταματήσω εδώ. Ό,τι είχα να πω το είπα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Μαρία. Πολύ δυνατό το μήνυμά σου τώρα. Η Σαρλότ πώς θα πάρει το λόγο. Well, it will be perhaps a bit more... Ίσως. Να είναι πιο δύσκολο. Ε, ε, αλλά νομίζω ότι πραγματικά έχω λάβει τέτοια έμπνευση και έχω τέτοιο ίστρο που θα είναι πολύ πιο εύκολο να κάνουμε ε, να επιτελέσουμε το έργο μας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, ευκαιρία που μας έδωσε να συμμετέχουμε σε μια τόσο σημαντική διάσκεψη και μέρα για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Σήμερα εορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα του Παιδιού και το μήνυμά μου προς εσάς είναι ένα απλούστατο μήνυμα. Σας παρακαλώ φροντίστε οι συζητήσεις ε, σε, στην καταπληκτική αυτή αίθουσα να ξεκινούν πάντα με το ερώτημα πώς αυτή η κατάσταση επηρεάζει τα παιδιά σήμερα, πώς θα επηρεάσει και τις μελλοντικέ γενιές. Και νομίζω ότι εκεί συμφωνούμε με τη Μαρία, γιατί η πιο σημαντική και βαρισίμαντη ερώτηση είναι ακριβώς αυτή. Φέτος, στην Παγκόσμια ημέρα του παιδιού, έχουμε την ευκαιρία να εορτάσουμε ένα σημαντικό ορόσημο, την 30η επέτειο της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Και όπως είπαν και πολλοί προλαλήσαντες, έχουμε την Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που έχει τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο ποσοστό κύρωσης από οποιαδήποτε άλλη συνθήκη. Από το 1989 η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει εμπνεύσει και έχει γίνει μοχλός σημαντικής προόδου για τα δικαιώματα των παιδιών. Όλο και περισσότερα παιδιά επιδώνουν τον πέμπτο γενεθλίο του. Όλο και περισσότερα παιδιά έχουν πρόσβαση σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και πολλέ αρχέ που κατοχυρώνονται και περιχαρακώνονται στη σύμβαση αυτή έχουν επηρεάσει εθνικά συντάγματα, ε, νομοθεσίε και πολιτικέ. Όπω η απαγόρευση των διακρίσεων, το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού, το δικαίωμα στη ζωή, στην επιβίωση, στην ανάπτυξη και το δικαίωμα στην προστασία. Και χαίρομαι ιδιαίτερω που η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και πάλι αποδεικνύεται παγκόσμιος ηγέτης ε, προκειμένου να μεταφέρει τα δικαιώματα των παιδιών σε προγράμματα, πολιτικές και υπηρεσίες που θα ωφελήσουν τις νεότερες γενιές και εντός και εκτός της Ευρώπης. Από το άρθρο 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας που προωθεί την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού ε, έως πολλές ε, νομοθετικές αλλαγές, πολιτικές και κατευθυντήρες γραμμές έχουμε μέσα και επενδύσεις που βελτιώνουν και προστατεύουν τα παιδιά παγκοσμίω. Έχουμε πολλές βελτιώσεις στο δικαστικό σύστημα προκειμένου να γίνει φυσικό προς, φιλικό προς τα παιδιά. Για παράδειγμα έχουμε τον συνήγορο του παιδιού στην Κροατία προκειμένου να συμπεριληφθεί ε, τα δικαιώματα του παιδιού. Επίσης στην Αυστρία έχουμε τα συμφέροντα του παιδιού, στη Σλοβενία Έχουμε τους φύλακες, τους επιμελητές για τους ε, ασυνόδευτους ανήλικες. Επίσης, έχουμε την ε, ιστορική διάλυση των συστημάτων ε, και χρηματοδότησης που έχουν ιδρυματοποιήσει τα παιδιά για πολλά χρόνια. Έχουμε όλο και περισσότερα παιδιά στη, σε, σε οικογενειακή φροντίδα ή στη φροντίδα της κοινότητας. 20 από τα 21 κράτη-μέλη έως τα 70 κράτη διεθνώς που έχουν ανανεώσει την δέσμευσή τους και έχουν κάνει νέες παγκόσμιες υποσχέσεις για την σύμβαση αυτή και μάλιστα η Ουκρανία ήταν η εκατοστή χώρα που το υποσχέθηκε. Πέραν τη πρόοδο που υλοποιήσαμε τι τρει τελευταίε δεκαετίε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και κάποιε αδυναμίε. Η μία που έχουμε υστερήσει. Στι χώρε ε, μεσαίου και χαμηλού εισοδήματο, τα παιδιά των φτωχότερων οικογενειών είναι, έχουν διπλάσια πιθανότητα να πεθάνουν από προβλέψιμε αιτίε πριν τα πέμπτα του γενέθλια από ότι ε, σε, τα παιδιά από πιο εύπορα νοικοκυριά. Και μάλιστα με βάση πρόσφατα στοιχεία, μόνο τα μισά παιδιά από τις φτωχότερες οικογένειες της Ποσαχάριας Αφρικής εμβολιάζονται για την ηλαρά σε σχέση με 85% των παιδιών των πλουσιότερων οικογενειών που εμβολιάζονται. Και παρά τη μείωση των, του ποσοστού των παιδικών γάμων, τα φτωχότερα κορίτσια σε κάποιες χώρες κινδυνεύουν πολύ περισσότερο σήμερα να τα παντρέψουν πρόωρα και καταναγκαστικά από ότι ε, το 1989. Τέτοιες προκλήσεις μάλιστα αντιμετωπίζουμε και εντός της Ευρώπης. Σήμερα ένα στα τέσσερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Μιλάμε δηλαδή για περίπου 25 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 18 ετών. Μερικέ φορές ακούμε νούμερα και δεν τα προσέχουμε, αλλά σκεφτείτε, 25 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω το 18 κινδυνεύουν με φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό. Παγκοσμίω, ένα στα τέσσερα παιδιά διαβιούν σε χώρες ε, που μαστίζονται από βίες ε, σειράξεις ή καταστροφές. 28 παιδιά απομακρύνονται από τα σπίτια τους λόγω της ανασφάλειας ή των πολέμων. Πολλά από τα παιδιά αυτά έρχονται σε ανεπτυγμένες χώρες, στην Ευρώπη αλλού, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά αυτό που βρίσκουν είναι σειρματοπλέγματα και τείχη ψηλά. Οπότε ο εορτασμό τη συνθήκη για τα δικαιώματα του παιδιού θα πρέπει να είναι και μια υπόσχεσή μα για το μέλλον. Μια δέσμευση των κυβερνήσεων να επενδύσουν σε όλα τα παιδιά. Γιατί αυτό είναι ηθική και πρακτική υποχρέωσή τους για να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Πώς θα επιταχύνουμε λοιπόν την πρόοδο. Καταρχάς, θα πρέπει να αφουγκραστούμε τα παιδιά και τους νέους το έχουμε πει. Η νέα γενιά γνωρίζει καλύτερα από οποιονδήποτε τι χρειάζεται. Κάθε χώρα λοιπόν θα πρέπει να διερωτηθεί πώς θα εμπλέξει καλύτερα τους νέους πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε προγράμματα και πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή των νέων. Αν οι κυβερνήσεις δεν προσφέρουν αυτό το, το παράθυρο διαλόγου στους νέους, οι νέοι θα το διεκδικήσουν τολμηρά και δυναμικά. Έχουμε δει εκατοντάδε χιλιάδε ε, νέων και εφήβων που κατέβηκαν στου δρόμου, διεκδικώντα το δικαίωμα σε ένα καθαρό και υγιή πλανήτη. Με άλλα λόγια, οι νέοι είναι έτοιμοι να γίνουν παράγοντε και φορεί αλλαγή. Αλλά η ερώτηση είναι, εμείς είμαστε έτοιμοι να το δεχτούμε. Όχι μόνο να τους ακούσουμε, αλλά να τους αφήσουμε να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο. Δεύτερον, Παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστήσει τα δικαιώματα του παιδιού πολιτική προτεραιότητα και εντό και εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε μια νέα φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού που θα μετατρέψει τις ε, πολιτικές δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα παιδιά σε ένα σχέδιο δράσης. Θέλουμε μια δέσμη συγκεκριμένων στόχων για τα παιδιά. Αυτά θα πρέπει να προσδιορίσουν το θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη πενταετία με συμμετοχή όλων των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών. Οι ευρωπαϊκέ πολιτικέ και κατευθυντήρε γραμμέ για τα δικαιώματα του παιδιού είναι μια καλή αφετηρία. Ένα σημαντικό επόμενο βήμα θα είναι να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπολογίσει τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών επενδύσεων στα παιδιά και να καταρτήσει μια ετήσια έκθεση με τα αποτελέσματα. Αυτό θα είναι μια σαφής απόδειξη της δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχουμε και καταμετρήσιμα αποτελέσματα αυτής της δέσμευσης. Τρίτον και τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό, καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη τις νέες ευκαιρίες και προκλήσεις για τα παιδιά. Μετανάστευση, κλιματική αλλαγή, ψηφιακές τεχνολογίες, επιθέσεις σε παιδιά σε σειράξεις και ψυχική υγεία. Πριν από 30 χρόνια αυτά τα θέματα δεν ήταν πρωτοσέλιδα. Η σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού δεν αναφερόταν συχνά. Όμω η σύμβαση αυτή περιλαμβάνει όλε τι αρχέ που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε αυτέ τι προκλήσει. Και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να είναι πρωτοπόρα και να βοηθήσει τα παιδιά ε, να αντιμετωπίσουν μαζί μας αυτές τις αλλαγές. Γιατί μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, πρωτοπόρα και πρωτοστάτησε σε, στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Θα πρέπει να συνεχίσει και να παραμείνει πρωταθλητής των δικαιωμάτων των παιδιών ευρωπαϊκά και παγκοσμίω. Και στο δρόμο αυτό η UNICEF θα είναι στο πλευρό σας, θα σας συμπαρασταθεί, θα είναι ο εταίρος σας, θα σας στηρίξει, ακόμη και θα σας παροτρύνει, θα σας παρακινήσει χώρες και νομοθέτες για να τηρήσετε όλοι τις υποσχέσεις που έχετε δώσει για τα παιδιά. Και το έργο που θα επιτελέσουμε σήμερα θα αποτελέσει το θεμέλιο για το μέλλον, για τα επόμενα 30 χρόνια. Και 30 χρόνια μετά ελπίζω να βλέπουμε το 2019 ως χρονιά όχι μόνο αναγνώρισης της σημασίας των δικαιωμάτων των παιδιών, αλλά και ως χρονιά που η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε κάτι για όλα αυτά. Ας μπούμε λοιπόν σε αυτό το ταξίδι μαζί με δυναμισμό και ενθουσιασμό. Ευχαριστώ. Θα δώσω μέσω στο λόγο στον Μπερεκέτ, ο οποίος είναι από την Αιθιοπία αλλά ζει στην Κάνα. Παρακαλώ, έχεις το λόγο. Όπω Όπως είπε ο προηγούμενος γενικός γραμματέας του ΙΕ, ο Μπάνκι μούν είπε λοιπόν ότι αυτό που έχουν κοινό όλα τα παιδιά είναι τα δικαιώματά τους. Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα στην επιβίωση, στην ανάπτυξη, παιδεία, στο να μην έχει να υποστεί βία και κακοποίηση και μπορεί να συμμετάσχει στην κοινωνία και να ακούγεται η φωνή του. Καλημέρα σας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να συμμετέχω στην 30η επέτειο εδώ τη ε, σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριουδάκι. Αντιουέλε λέγεται και βρίσκεται στην περιοχή Μεκέλε στη Βόρεια Αιθιοπία. Λέμε στα αμχαρικά ότι ένα παιδί πρέπει πάντοτε να έχει την τύχη να μεγαλώσει. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται πάντα. θα πρέπει να έχουν όλοι οι γονείς την κατάλληλη στάση όσον αφορά τα παιδιά ε, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να τα μεγαλώσουν, δεν μπορούν να τους δώσουν ε, το φαγητό. Πολλές φορές δεν αφιερώνουν χρόνο και χρήμα στα παιδιά τους και αφήνουν τα παιδιά στην τύχη τους. Τα περισσότερα παιδιά στην Αιθιοπία αρχίζουν να δουλεύουν ε, στο αγρόκτημα, στο χωράφι του μπαμπά τους μόλις τα τέσσερα και πολλοί πρέπει να αρχίσουν το σχολείο. Και 33% των παιδιών στην Ήπεθρο περπατάνε πάνω από 5 χιλιόμετρα για να πάνε στο σχολείο. Σε τρομερές συνθήκες πρέπει ε, να κάτσουν για να διαβάσουν κάτω από τα τρένα και θα πρέπει να διαβάσουν με άδειο το στομάχι. Θα πρέπει να πασχίσουν μέρα και νύχτα για να βρουν τελικά κάποια στιγμή το φαγητό που θα τους εξασφαλίσει την ανάπτυξη. 61,8 των παιδιών στην ε, Ήπεθρο εγκατελείπουν το σχολείο. Και το μέλλον των ε, αγοριών είναι να γίνουν ε, γεωργοί και των κοριτσιών να γίνουν μητέρες. Εγώ είχα την τύχη να ακολουθήσω ένα διαφορετικό δρόμο χάρη ε, στα SOS, ε, τα χωριά, τα παιδικά SOS, Children Village. Και είχα μια ανάδοχη οικογένεια που με αγαπούσε πολύ και είχαμε ένα σχολείο με πλούσια βιβλιοθήκη έγινα μέλος του Κοινοβουλίου των Παιδιών εκπροσωπώντα το χωριό μου και μετά έγινα πρόεδρο αυτού του κοινοβουλίου. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Έτσι μπόρεσα να φροντίσω του ομοίου μου, τι ανάγκε τους και κάποια στιγμή ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα για να μπορέσουμε να γιορτάσουμε το νέο έτος με μη προνομίουχα παιδιά εκτός των παιδικών χωριών. Περάσαμε τη μέρα μαζί ε, τους, προσφέραμε φαγητό. Αυτό τώρα έγινε μια ετήσια εκδήλωση. Και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου ήταν όταν πήρα μια υποτροφία για να πάω ε, σε ένα πάρα πολύ έγκυρο φημισμένο ε, σχολείο πανεπιστήμιο στην Κάνα. Όλα αυτά γιατί σας τα λέω, γιατί σας λέω ότι ζωή μου. Γιατί γίνονται κάποια πράγματα θαυμαστά όταν υπάρχει σεβασμός για τα παιδιά, προστασία για τα παιδιά, βοήθεια προς αυτά. Και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει εγώ να είμαι η εξαίρεση. Ονειρεύομαι. Μια μέρα να βοηθήσω να αλλάξει η ζωή των παιδιών. Και θα το λέω γιατί θεωρώ ότι αυτό δεν κοστίζει πολύ μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής τους και όλοι να μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο αυτό θα αλλάξει τη ζωή τους, το μέλλον τους το μόνο το οποίο χρειάζεται να κάτσει το παιδί στο σχολείο είναι το να έχει σωστή διατροφή οπότε όλοι μαζί ας προσπαθήσουμε η ζωή εκατομμύριων παιδιών στη ζωή μου και παντού στον κόσμο να είναι έτσι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπερεκέτ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, ε, Βελίνα τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Παιδιού στα Ηνωμένα Έθνη. Ε, σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, παιδιά, συνάδελφοι, μεγάλη μου τιμή η ευκαιρία που έχω να γιορτάσω μαζί σας την επέτειο αυτή ως μέλος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ως Ευρωπαία Πολίτης. Η Επιτροπή μας είναι το όργανο που ορίζει η σύμβαση ε, για να παρακολουθεί την εφαρμογή της και την υλοποίησή της. Η Επιτροπή αυτή συνεδριάζει, συναντάει κυβερνήσεις αλλά και παιδιά τρεις φορές το χρόνο στη Γενέβη και με την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις της, ε, τους διαμεσολαβητές, τους συνήγορους του παιδιού, για να συλλέγει περισσότερες προφορίες για την κατάσταση των παιδιών σε κάθε χώρα. Η Επιτροπή μας λοιπόν είναι η κατεξοχήν αρμόδια για να γνωρίζει τι γίνεται και πώς εφαρμόζεται παγκοσμίω η σύμβαση αυτή. Έχω προετοιμάσει μια γραπτή ομιλία την οποία δεν πρόκειται να διαβάσω μετά από μισή μέρα συζητήσεων για τη σύμβαση. Θα ήθελα όμως να τονίσω τα εξή δύο. Τι γιορτάζουμε ακριβώς σήμερα και τι θα ε, πρέπει να περιμένουμε ε, από το μέλλον, στα επόμενα 30 χρόνια ας πούμε. Η Επιτροπή μας θα μπορούσε να σας απαντήσει το εξής. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η έγκριση της σύμβασης αυτής πριν από 30 χρόνια ορίστηκε ως νομική και ε, πολιτισμική επανάσταση. Γιατί νομική. Γεννήθηκε διεθνές δίκαιο που θα δώσει, έδινε δικαιώματα στα παιδιά σε ίσο επίπεδο με τους ενήλικους. Αλλά και πολιτισμική επανάσταση γιατί ε, αυτό σήμαινε ότι αλλάζουν οι κανόνες, τα ε, στερεότυπα για τα παιδιά που είχαν δημιουργηθεί εδώ και αιώνες και βασίζονταν σε εξουσίες και δομές, είτε αυτές είναι κοινωνικές, οικογενειακές κλπ. Αυτή ήταν η βασική φιλοδοξία της σύμβασης. Είναι να αλλάξει το παιχνίδι των εξουσιών νομική επανάσταση κανονικά θα ερχόταν να υποστηρίξει και την πολιτισμική αλλαγή που επρόκειτο να κάνει πραγματικότητα τα δικαιώματα για όλα τα παιδιά. Τότε είχε γεννηθεί μια ελπίδα ότι η δέσμευση που γρήγορα έδειξαν ε, ε, όλοι ε, και η καθολική αποδοχή θα σήμαινε αποτελέσματα, με πολιτικές, με ηγετική στάση για να αλλάξουν αυτές οι πεπιθήσεις, οι νοοτροπίες αλλά και η ζωή των παιδιών. Και μάλιστα ήταν πολύ σημαντικό αυτό, ήταν χειρό και το μήνυμα το οποίο παραμένει ότι τα παιδιά θα πρέπει να ε, ε, χειραφετηθούν και να έχουν την υποστήριξη και τις δυνατότητες να συμμετέχουν, να εισακούονται όπως κάθε ε, άνθρωπος και κάθε άνθρωπος που έχει δικαιώματα. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους μας ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θεμέλιο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Και η προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και αφορά τα παιδιά θα πρέπει να είναι τμήμα τη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά στην πρωτοπορία της παγκόσμιας ατζέντα και ποτέ δεν το ξεχνάμε. Τα δικαιώματα των παιδιών ε, έχουν κατοχυρωθεί στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο, αλλά και στην ομολογία των δύο διεθνών δικαστηρίων στην Ευρώπη. Τα παιδιά είναι ψηλά στις προτεραιότητες πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που εφαρμόζονται όχι μόνο στην Ένωση αλλά και διεθνώς. Αυτά είναι λοιπόν τα επιτεύγματα που σήμερα γιορτάζουμε. Ωστόσο... Οι καλές πρακτικές και η καλή νομοθεσία δεν έχει φτάσει σε όλα τα παιδιά όπως ακούσαμε σήμερα ε, πάρα πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα. Εκτός από τη φτώχεια, η ιδρυματοποίηση, η βία και η σωματική τιμωρία παραμένουν αποδεκτές μέθοδοι πιθαναγκασμού των παιδιών στην Ευρώπη. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναγνωρίζει ε, κάποια επίγοντα θέματα. Ε, μιλήσαμε για την κλιματική αλλαγή παγκοσμίω, μιλήσαμε για τις δραστηριότητες ε, της οικονομίας που επηρεάζουν αρνητικά τα δικαιώματα των παιδιών. Αναφερθήκατε προηγουμένως στο γάλα στην Αφρική. Επίσης, συζητήσαμε άλλα θέματα, όχι τη διαφθορά, τις ένοπλες σειράξεις, τις πολιτικές αστάθειες, την άνοδο του εξτρεμισμού και την αυξανόμενη οικονομική ε, παγκόσμια ανισότητα. Όλα αυτά τα θέματα είναι επιζήμια για τα δικαιώματα των παιδιών και δεν θα πρέπει ποτέ να τα ξεχνάμε. Και ελπίζω το νέο κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη αυτά τα θέματα και προσβλέπουμε σε αυτό. Οι επέτειοι και τα γενέθλια ε, συνδυάζονται με ευχές και με δώρα για το μέλλον. Ποιες είναι οι ευχές μας για τα σημερινά και τα αυριανά παιδιά. Ίσως θα μπορούσαμε αυτές τις ευχές να τις συνδέσουμε με ε, την ε, φιλόδοξη ατζέντα για το 2030 που έχουμε συμφωνήσει παγκοσμίω. Θα ήθελα επίσης να τονίσω κάτι ακόμα. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού φρονεί ότι η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και με ισότητα παγκοσμίω δεν μπορεί ε, να γίνει χωρίς να είναι τα παιδιά ενεργοί ε, συμμετέχοντες και πρωταγωνιστές σε αυτή την προσπάθεια. Πολύ πρόσφατα έγινε μια μελέτη στην Ευρώπη που αποκάλυψε μεταξύ 20.000 παιδιών έγινε αυτή η μελέτη στην Ευρώπη. Αποκάλυψε λοιπόν ότι μόλις το 15% των παιδιών στην Ευρώπη αισθάνονται ότι ακούν τη γνώμη τους οι ενήλικοι όταν παίρνουν τις αποφάσεις και λιγότερο 8% θεωρούν ότι λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις τους όταν παίρνονται αποφάσεις στην κοινωνία. Υπάρχει ένα πρωτόκολλο προαιρετικό ε, στη Σύμβαση το 2011 για τις διαδικασίες επικοινωνίας θα ήθελα να το γνωρίζετε και εσείς και τα παιδιά. Το πρωτόκολλο αυτό μέχρι στιγμής έχει κυρωθεί από 46 κράτη συμβαλόμενα μέρη της σύμβασης τα οποία είναι 196. Μόλις 46 από τα 196 κράτη, εκ των οποίων μόλις 14 είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ας καλέσουμε από κοινού όλα τα ευρωπαϊκά κράτη τουλάχιστον να υπογράψουν αυτό το προαιρετικό πρωτόκολλο που είναι ακόμα ένα μέσο και εργαλείο για να επιταχυθεί η υλοποίηση ε, της σύμβασης και η συμμετοχή των παιδιών. Αυτά. Και τελευταίο, η 30η επέτειος της σύμβασής μας μας δίνει μια νέα όθηση για ανανέωση της δέσμευσης των κυβερνήσεων υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών. Τα ακούσαμε αυτά προηγουμένως. Hopefully. Hopefully. Ελπίζω και επειδή είναι αφιερωμένο το πάνελ στα όνειρα, ελπίζω να μπορούμε να ονειρευτούμε ότι μετά από 30 χρόνια θα ξανάρθουμε και πολλές κυβερνήσεις θα είναι περήφανες που θα έχουν υλοποιήσει όλα αυτά τα όνειρα και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν για τα δικαιώματα των παιδιών. Ευχαριστώ. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο ε, ε, στο κοινό. Έχετε ζητήσει πάρα πολύ το λόγο και θα είμαι αυστηρή. Ε, λιγότερο αυστηρή με τους νέους. Λιγότερο νέοι θα έχετε ένα λεπτό. Τώρα θα κάνω διάκριση εγώ υπέρ των νέων. Φαμπιέν Βαντενέντε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, από την ΤΕΦΚΟ, από το Τμήμα ε, Ανθρώπινα Δικαιώματα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όχι, δεν είμαι από τους πολύ νέους, άρα θα έχω μόνο ένα λεπτό εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ, Ανάπτυξη Συνεργασία, εμπνευσμένες οι ομιλίες ιδίως από τους δύο νέους ηγέτες και αναφέρθηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είμαστε πρωτοπόροι όσον αφορά τα δικαιώματα των ανηλίκων και ότι δεσμευτεί να το κάνει αυτό η νέα Επιτροπή. Να σας πω τι κάνουμε και τι θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θέλουμε να φρενάρουμε την βία κατά κοριτσιών και γυναικών Οκτώ χώρες στην Αφρική, πέντε στη Λατινική Αμερική. Υπάρχει μια συνεργασία ε, και συνεργαζόμαστε με πολιτικούς, κυβέρνηση για των πολιτών. Θέλουμε να είναι η παιδεία ε, φιλική στα παιδιά, να υπάρχει σύστημα προστασίας και για την βία. Έχουμε τη χρηματοδότηση. Και τελειώνω, τελειώνω τώρα. Απλώς να σας πω ότι μέχρι τώρα 64 εκατομμύρια έχουν διατεθεί για αυτή μας την ε, πολιτική κατά της βίας. Σας ευχαριστώ. Και τώρα τον λόγο έχει η Μαριάν Έριξον, ε, διευθύντρια της ε, οργάνωσης Διεθνέ πλάνο τη Σουηδίας. Πάρα πολύ εμπνευσμένα όλα αυτά μας είπαν είναι εδώ όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι μας δίνουν ελπία η ευφία τους και αφού γκράζουμε τους νέους που ξέρουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό είναι θέμα σημαντικό για την ε, σύμβαση των δικαιωμάτων. Να ξέρουμε λοιπόν μας ότι κάποια πράγματα έχουν εκτροχιαστεί. Τι μας λένε οι νέοι, ότι θέλουν η Ένωση να είναι ο ενήλικας να λάβει τις ε, αποφάσεις κατάλληλη νομοθεσία, κατάλληλη προοικοδότηση θέλουν να σταματήσουν και τροχιασμό τα πράγματα να ξαναπάρουν την ε, ρότα τους για έναν καλύτερο, πιο δίκαιο κόσμο. Και κανείς να μην χάνει αυτό το τρένο. Η Μαρία Λόντερ, συντονίστρια για τα δικαιώματα του παιδιού στο Global Campus για τα δικαιώματα του παιδιού. Thank you very much for the opportunity. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Είμαι ε, συντονίστρια για τα δικαιώματα του παιδιού στο Global Campus Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι μεταξύ ε, εκπαίδευσης, έρευνας και ακτιβισμού και συμβάλλουμε, ε, στην εκπόνηση της έκθεσης που δημοσιεύθηκε χθε στην Γενέβη. Και φυσικά στο πάνελ αυτό με θέμα κάθε παιδί ε, έχει δικαίωμα στο όνειρο. Τα παιδιά που έχουν στερηθεί την ελευθερία τους φυσικά δεν έχουν κανένα δικαίωμα στο όνειρο. Γιατί όταν στερούμε από τα παιδιά την ελευθερία τους, στερούμε την παιδική τους ηλικία. Και σε αυτή την ε, μελέτη 273 ε, παιδιά συμμετείχαν ενεργά, ε, παρουσίασαν την ιστορία τους, ε, υπέστησαν προβλήματα λόγω μετανάστευσης, σειράξεων, εθνικής ανασφάλειας, ιδρυματοποιήθηκαν πάνω από 7 εκατομμύρια παιδιά στερήθηκαν την ελευθερία τους. Και η ερώτησή μου εδώ προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που συνέβαλε σημαντικά στην εκπόνηση της μελέτης αυτής όπως και η UNICEF είναι τι μπορούμε να κάνουμε ώστε οι συστάσεις ε, να περάσουν σε έμπρακτες ε, ε, ενέργειες και κανένα παιδί να μην υποστεί κράτηση επειδή απέτυχαν τα συστήματα που εκπώνησαν οι ενήλικες. Φρανσουά Ντεμπέρκτ, απεσταλμένος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και των νέων. Συγγνώμη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση που είναι απλούστατη και πολύ σύντομη. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε εδώ ότι οι νέοι έχουν δικαίωμα να εκφέρουν τη γνώμη τους και να εισακουστούν. Όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Και όμω, συμφωνώ με τη διαπίστωση τη κυρία Τοντόραβα. Γιατί ένα μεγάλο τμήμα των νέων έχουν ακόμη την αίσθηση ότι η φωνή τους δεν ακούγεται και δεν φτάνει εκεί που θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη, δηλαδή εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Και είναι ρητορική αυτή η ερώτηση, γιατί σήμερα διαπιστώνουμε ότι στους τομείς που μπορεί πραγματικά να σημειώσουμε πρόοδο. Εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για παράδειγμα, και στην κοινωνία, η φωνή των νέων δεν λαμβάνεται δεόντως υπόψη. Θα ζητώ λοιπόν επίσημα να εφαρμόσετε το συντομότερο δυνατό κάποιους, κάποιους νομοθετικές θεσμικές διάβλους, ώστε να, να εξασφαλίσετε την ανάμεξη και των νέων, όπως το Φόρουμ των ε, Νέων Κοινοβουλευτικών, για να έχετε και την άποψη των νέων ε, και τη δική τους γνώμη για, το, για τις αποφάσεις ε, που θα διαμορφώσουν το μέλλον τους και το μέλλον μας. Η Ειρήνα Φομβίσοκ που είναι Ευρωβουλευτής και μέλος Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Είμαι Βρετανίδα που είναι σίγουρα από τις πιο εύπορες ε, και τυχερές κοινωνίες του κόσμου. Και φυσικά αυτό που θα πω εγώ δεν επισκιάζει τη σημασία των προβλημάτων που επισημάθηκαν. Ακόμη όμως και στη δική μου πατρίδα, περιπτώσεις ε, ψυχικών προβλημάτων παιδιών ε, αυξάνονται. Οι νέοι σήμερα νιώθουν ε, μεγάλη ένταση και πίεση. Η μεγάλη μου κόρη που είναι 15 χρονών λέει ότι δεν θέλει να ακολουθήσει τα βήματά μου και να γίνει πολιτικός γιατί βλέπει τι κακομεταχείριση δέχομαι διαδικτυακά και φυσικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνέβαλαν σε αυτήν την κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν τα θέματα ψυχικής υγείας να αντιμετωπίζονται εξίσου σοβαρά με τα θέματα σωματικής υγείας για τους νέους. Θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα και να αλλάξουμε το δημόσιο μας αφήγημα, να το κάνουμε πιο πολιτισμένο και πραγματικά να ανταποκρίνεται στην οριμότητα που θα πρέπει να δείχνουν οι ενήλικες. Ευχαριστώ. Um, Εγώ είμαι μέλος της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων Γυναικών και Ισότητας ε, στο Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό και είχα την ευκαιρία να είμαι στον Ναϊρόμπι την περασμένη εβδομάδα στη Διεθνή Διάσκεψη για την Ανάπτυξη και τον Πληθυσμό και κατάλαβα ξεκάθαρα ότι ε, αν θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτά που λέει ο χάρτης ότι κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται θα πρέπει να χειραφετήσουμε τις γυναίκες περισσότερο από οτιδήποτε, ιδιαίτερα τις νεαρές γυναίκες. Και έχω ένα μήνυμα προς τους άνδρες εδώ, ότι θα πρέπει εμείς να αγωνιστούμε για την ισότητα των φύλων. Αυτό δεν μπορεί να αφαιθεί στα χέρια των μισών ανθρώπων, να αγωνίζονται γυναίκες για τα γυναικόματά τους. Γιατί αν οι γυναίκες καταφέρουν να ονειρεύονται, αυτό θα είναι καλό για την κοινωνία. Και το λέω και προς τους νέους. Ε, ε, στα νεαρά αγόρια ότι έχετε κι εσείς ρόλο να παίξετε. Γυρίστε πίσω και βοηθήστε κάθε παιδί να υλοποιήσει τα δικαιώματα και τα όνειρά του. Ευχαριστώ. Alors, on a une demande de... Η νόμη Ισαμπέλα από την Ομβέρσα ζητεί το λόγο. Μαθήτρια Λυκείου. Μαθήτρια Λυκείου. Σήμερα γιορτάζουμε αυτήν την Σύνοδο Υψηλού Επίπεδου για την 30η επέτειο της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Σας ευχαριστούμε για αυτή την εκδήλωση και που μας καλέσατε. Το 1989 είναι γιατί απίστευτο. Οι αρχηγοί και οι ηγέτες έφτιαξαν αυτήν την ε, συνθήκη και υποσχέθηκαν ότι κάθε παιδί θα μπορεί να έχει τα δικαιώματά του αυτό το οποίο σήμερα γιορτάζουμε. Και εγώ όπως και τα άλλα παιδιά είμαστε ευγνώμονες που έχουμε αυτά τα δικαιώματα και ότι έχουμε το δικαίωμα στη γνώμη μας. Όπως το είπαν και οι προηγούμενοι. Αυτό είναι απίστευτο. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ακόμα έχουμε δουλειά μπροστά μας. 186 εκατομμύρια παιδιά έχουν χάσει την παιδική του ηλικία γιατί πρέπει να δουλεύουν. Πάνω από 150 εκατομμύρια παιδιά εκτίθενται σε κινδύνους, νάρκες κλπ. Οπότε θα πρέπει να δουλέψουμε για το μέλλον αυτών των παιδιών να μπορούν να έχουν τα δικαιώματά τους. έχουμε ένα ίδρυμα που έχει ως έργο τη βοήθεια της Αφρικής παιδεία για τα παιδιά και για τους νέους. Βοηθούμε το Κονγκό, το μέλλον των παιδιών, εκεί. Ούτως ώστε να συνεργαστούμε με, για τέτοια προγράμματα. Και το Ίδρυμά μας σας ευχαριστεί επίσης. Μπεντσαλή ε, στο έδρο 64. Ναι. Σας ευχαριστώ καταρχάς κυρία Πρόεδρε. Στη συνέχεια θα ήθελα να σας ζητήσω, να σας ρωτήσω όλους ε, ξέρετε τι σημαίνει πείνα. Δεν λέω αυτό το αίσθημα της πείνας που νιώθω τώρα, επειδή πεινάω, αλλά μιλάω για ένα αίσθημα που σε παραλύει, που δεν ε, σε αφήνει να σκέφτεσαι το σχολείο, του ερωτέ σου. Λέγομαι Ουσάμα, είμαι 19 ετών. Εγώ δεν ξέρω τι σημαίνει να πεινάς. Και σε ευχαριστώ, Μπερικέτη, για αυτά που είπες. Θα ήθελα να σας μιλήσω για αυτά τα παιδιά που δεν έχουν τη δική μου τύχη, που δεν έχουν τη δική μας τύχη. Ιδιαίτερα εδώ μιλώ για τα παιδιά της Ιεμένης που ε, εφίστανται τον πόλεμο που έχουν ε, αποφασίσει οι ενήλικες και μετά εφίστανται και την πείνα. Κάθε μέρα βομβαρδίζει εκεί η Σαουδική Αραβία και οι σύμμαχοί της. Ξέρω ότι είναι σημαντικό να διατηρήσεις ένα πολιτικό και οικονομικό σύμμαχο και εταίρο, αλλά δεν αρκεί αυτό απέναντι στα δεινά που προκαλούν ε, στους νέους και τα παιδιά. Με το ένα χέρι ε, πουλάμε όπλα στη Σαουδική Αραβία και με το άλλο μετράμε τους θανάτους και ε, κλεγόμαστε. Τι υποκρισία αυτή. Ζητώ όπως και η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να πουλάει όπλα στη Σαουδική Αραβία. Δώστε μου μία ευκαιρία τουλάχιστον να είμαι περήφανος που είμαι Ευρωπαίος. J'espère qu'on en offrira plus qu'une. <laughs> Euh, Ελπίζω να σας δώσουμε πάνω από μία. Η κυρία Κασαλκό, στην, στο έδρανο υπαριθμών 6. Γεια σας. Είμαι παιδί από διαφορετικές κουλτούρες. Η αδικία και η δυστυχία Ε, προέρχονται από διαφορετικούς λόγους. Ενώ η ευτυχία και οι ευτυχείς κοινότητες έχουν ε, κοινούς και ισχυρούς πυλώνες. Μετά από μία ημέρα που ακούσαμε πολλές ομιλίες, θα ήθελα να σας ζητήσω το εξής. Ένα συγκεκριμένο σχέδιο και σαφείς στόχους και ε, εκτέλεση, εφαρμογή του σχεδίου που θα αξιολογείτε και θα παρακολουθείτε. Ευχαριστώ. Παλιέρο Ζωζέ, στη θέση 147. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, νιώθω μεγάλη τιμή που συμμετέχω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους και λαμβάνω το λόγο εδώ. Εδώ και 18 χρόνια είμαι καθηγητής, ε, δάσκαλος μάλλον πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εδώ εορτάζουμε τη σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο άρθρο 9 που λέει ότι σε καμία περίπτωση ένα παιδί θα πρέπει να χωρίζεται από τους γονείς του. Βέβαια, στην Ισπανία, στις δίκες διαζυγίου, δεν δίνονται όλες οι δικονομικές εγγύησεις και οι γονείς στερούνται το ανθρώπινο δικαίωμά τους ε, του τεκμηριωθότητας και δεκάδες χιλιάδες παιδιά στην Ισπανία δεν μπορούν να είναι με τους γονείς τους εξαιτίας ε, των χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών και των χρονοβόρων δικών. Και επίσης ε, δεν μπορούν να απολαύσουν ούτε την συντροφιά των παππούδων τους. Έχω δύο παιδιά και τον επόμενο μήνα, τα Χριστούγεννα, θα είναι τα πέμπτα Χριστούγεννα που δεν θα μπορώ να είμαι με τα παιδιά μου. Ε, ενώ το ισπανική κυβέρνηση μου επιτρέπει να, να μορφώσω τα παιδιά των άλλων, δεν ε, με, μου επιτρέπουν να διαπαιδαγωγήσω τα δικά μου παιδιά. Και τέτοιες περιστάσεις έχουμε σε δεκάδες χιλιάδες διαδικασίες διαζυγίου, στις οποίες δεν δίνονται οι απαραίτητες δικονομικές εγγυήσεις. Δεν εφαρμόζεται το άρθρο 9. Και επειδή η μαμά μου, η γιαγιά που θα μπορούσε να κάνει μελομακάρονα για τα παιδιά, για τα γονάκια της αυτά τα Χριστούγεννα, δεν έχει αυτή την ευκαιρία και σε ζητώ βοήθεια εκ μέρους δεκάδων χιλιάδων γονιών από την Ισπανία, πατέρων. Θα δώσω το λόγο στον τελευταίο ομιλητή, στη Φάραο Κάση, στο 232. Hello everyone. Γεια σας. Σας ευχαριστώ όλους για τις απόψεις σας. Πραγματικά φωτίζετε διάφορες πτυχές και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, για να τονίσω κι εγώ κάτι. Όταν ήμουν πιο μικρή ήμουν αυτιστική. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Σουηδία. Οι γονείς μου κατάγονται από το Μαρόκο και είχα την τύχη να έχω αυτό το κράτος πρόνοιας που με υποστήριξε. Σήμερα είμαι αυτή που είμαι. Και θα ήθελα να πω ότι είναι πολλά τα παιδιά, ακόμα και στην Σουηδία, με ξένη καταγωγή που δεν πιστεύουν στα όνειρά τους. Και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Στη Σουηδία ως παιδί μπορεί να έχεις μια καλή ζωή εντός εισαγωγικών και να μεγαλώσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η κοινωνία δεν αποκλείει κάποια παιδιά. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι πρέπει όλοι να πιστεύουμε σε όλα τα παιδιά πάντα. Και κάθε παιδί έχει διαφορετική σκοπιά από την οποία το βλέπει για να μπορέσει να ανθίσει και να μεγαλώσει, όπως και εγώ. Αυτό ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την οπτική του καθενός και συνεχίστε την καλή δουλειά που κάνετε. Ευχαριστώ. Euh, σας ευχαριστώ πολύ για όλες σας τις παρεμβάσεις. Δεν θα απαντήσουμε σε όλες τώρα, αλλά να είστε βέβαιοι ότι όσα είπατε θα συμπεριληφθεί στις εργασίες που έχουμε ο κάθε βουλευτής στην κάθε επιτροπή μας. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να ασχολούμαστε με τα ε, δικαιώματα του παιδιού σε μία επιτροπή, στη δική μας υποεπιτροπή, αλλά σε όλες τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των άλλων θεσμικών οργάνων. Όλα είναι άλλωστε αλληλένδετα και να είστε βέβαιοι ότι οι προτάσεις που κάνατε θα έχουν συνέχεια και οι προτάσεις που έκαναν οι οργανισμοί που σας εκπροσωπούν συχνά. Μας εμπιστεύονται ε, κάποια αποστολή. Ε, θα δώσω το λόγο τώρα στην κυρία Κέμπα που θα μιλήσει εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, αλλά και πολύ αγαπημένα παιδιά και νέοι. Ε, θα πρέπει να κλείσω κάποια συμπεράσματα από αυτό το πάνελ που είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί μιλά για το το δικαίωμα των παιδιών, το δικαίωμα στο όνειρο. Αυτό είναι αναφέρετο και αναπαλωτρίο το δικαίωμα, το δικαίωμα στο όνειρο. Ε, έχετε δικαίωμα στο όνειρο, το όνειρο άλλωστε είναι και ο μοχλός των δράσεών μας. Και μάλιστα όλοι οι νέοι, όλα τα παιδιά που πολλές φορές βρίσκονται σε πολύ δύσκολη τραγική κατάσταση ε, νομίζω ότι και τα δικά του όνειρα αντίχησαν εδώ και σας είμαι ευγνώμων ιδιαίτερα εμείς ε, οι θύνοντες πολιτικής που θα έχουμε επιρροή σε πολλές αποφάσεις που λαμβάνονται και στις πατρίδες μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χαίρομαι που οργανώσαμε αυτή τη διάσκεψη. Το παιδί, τα παιδιά ε, είναι η πιο ευάλωτη ομάδα της κοινωνίας γιατί είναι η πιο ανυπεράσπιστη ομάδα, είναι ανήμπορη ομάδα και θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να υλοποιήσει το, τα όνειρά τη αυτή η ομάδα και αυτό είναι καθήκον να εξασφαλίσει αυτή την υλοποίηση του ονείρου είναι καθήκον των ενηλίκων. Ακούσαμε τα όνειρά σα, ακούσαμε ε, για τα δικαιώματα των παιδιών. Έχουν περάσει 30 χρόνια από την υιοθέτηση τη συνθήκη και παρόλα αυτά η συζήτηση εξακολουθεί να είναι επίκαιρη και σε μερικέ περιοχές του κόσμου είναι ακόμη πιο επίκαιρη, εξαρτάται από την κατάσταση. Αλλά πρώτα απ' όλα ακούσαμε αυτά που μας είπε η Μαρία από το Σουδάν, το δικαίωμα των παιδιών να μην είναι θύματα βίας. Αυτό είναι θεμελιώδες δικαίωμα και θα πρέπει να το προστατεύσουμε και να το διαφυλάξουμε. Αν δεν μπορεί να το καταφέρει ε, ένα κράτος, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διεθνή συνεργασία και το διεθνές δίκαιο και να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί. Επίσης, ακούσαμε το δικαίωμα των παιδιών αλλά και των ανηλίκων σε καθαρό περιβάλλον, σε καθαρό αέρα. Θα πρέπει λοιπόν οι θύνοντες πολιτικές να λάβουν υπόψη όλα αυτά τα θέματα. Επίσης το δικαίωμα στην παιδεία, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, το όνειρο για το σχολείο, το δικαίωμα για το όνειρο για τις σπουδές. Αυτό μας είπε ο φίλος μας ο Μπερέκετ. Ένα δολάριο, ένα δολάριο αρκεί για να εξασφαλίσει την πρόσβαση ενός παιδιού στο σχολείο. Αυτό είναι αδιανόητο για τις πλούσιες χώρες πιο εύπορες, όμως αυτό συμβαίνει και θα πρέπει να το φροντίσουμε. Το δικαίωμα στην ασφάλεια επίσης. Το δικαίωμα του παιδιού είναι το δικαίωμα του ανθρώπου, όπως μας είπε και η Μαρία. Θα πρέπει να βοηθήσουμε επίσης τα θύματα της βίας. Και επίσης το δικαίωμα στην ε, ιατρική περίθαλψη, άσχετα με το κοινωνικό καθεστώς, άσχετα με την κοινωνική θέση. Γιατί αυτό είναι το όνειρο του παιδιού, να έχει πρόσβαση στην υγεία και όχι μόνο τα παιδιά εύπορων οικογενειών να έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη. Ακόμη και τα παιδιά οικογενειών χαμηλού εισοδήματος να έχουν πρόσβαση στην υγεία. Επίσης θα πρέπει να συνενώσουμε τις προσπάθειές μας όλοι, όλα τα θεσμικά όργανα και η σημερινή συνέλευση που είναι πραγματικά μια ε, πολύ καλή έκκληση και προσπάθεια για την λήψη υπόψη της ε, άποψης των παιδιών. Και επίση το πιο σημαντικό αίτημα και πιο σημαντική έκκληση είναι η έκκληση για την ειρήνη. Αυτό είναι ένα μήνυμα που στέλνουμε προ του διπλωμάτε όλου του κόσμου, γιατί τα παιδιά είναι αυτά που πλήττονται περισσότερο από τις ένοπλες σειράξεις. Αυτά είναι τα πρώτα θύματα των ένοπλων σειράξεων και θα ήθελα να ευχαριστήσω οργανώσεις όπως τη UNICEF. Ε, ως υπουργό ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια συνεργάστηκα με την UNICEF και ε, ο Γιάννος Κόρτσακ, ο επιφανής Πολωνός που έδωσε ε, μάχη για τα δικαιώματα του παιδιού. Και θα ήθελα να πω στη Μαρία από την Ουγκάντα ότι πήγα στην Ουγκάντα στο μεγαλύτερο καταβλισμό προσφύγων σε μια χώρα που σπαράζεται από το πόλεμο και 71% ε, των παιδιών ε, των, των διαμενόντων στον καταβλισμό ήταν παιδιά, παιδιά που πέθαιναν στην αγκαλιά μου. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε οργανώσεις όπως η UNICEF, η UNICEF να στηρίξουμε μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τους νεαρούς εθελοντές, γιατί εσείς οργανώνεστε. Γιατί στην Ιορδανία έχουμε νεαρούς ε, εθελοντές από τη UNICEF. Ε, έπεισαν ε, τους γονείς να στείλουν τα παιδιά στο σχολείο. Και χάρη σε αυτή την προσπάθεια πολλά παιδιά κατάφεραν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Και μου είπαν πολύ επιτρέψτε μας να ανακτήσουμε την αξιοπρέπειά μας, να, να καλλιεργήσουμε τις ε, ικανότητές μας, τις δεξιότητές μας, να ξεπεράσουμε το πόλεμο. Θέλουμε να επιστρέψουμε στις αιστείες μας, να ξαναφτιάξουμε τα σπίτια μας. Και χάρη στην συνεργασία με τη UNICEF ε, ε, χρηματοδοτήσαμε ένα επαγγελματικό λύκειο. Από κοινού πολλά μπορούμε να κάνουμε και έχουμε πραγματικά ένα ιερό καθήκον να υλοποιήσουμε αυτά τα όνειρα των παιδιών και των νέων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται το πάνελ και θα δώσω αμέσως το λόγο στην Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κυρία Κόπατς. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί νέοι, αγαπητά παιδιά, θα ήθελα να κάνω μια ανακεφαλαίωση της σημερινής διάσκεψης. Πριν όμως ε, κάνω μια σύνοψη της σημερινής ημέρας, θα ήθελα να κάνω μια δήλωση. Εδώ και ε, τρεις μήνες είμαι Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά εδώ και για πολλά χρόνια ήμουν γιατρός και ασχολήθηκα με την θεραπεία παιδιών και το σημαντικότερο που έμαθα είναι να ακούω τα παιδιά κατά την μακρά μου σταδιοδρομία ως παιδίατρος και είναι πραγματική δεξιότητα να μπορεί κανείς να ακούει και αυτή την δεξιότητα θα τη χρησιμοποιήσω στο αξίωμα που έχω τώρα ως συντονίστρια για τα δικαιώματα των παιδιών. Θα ακούσω τη φωνή των παιδιών και των νέων και είμαι στη διάθεσή σας, στη διάθεση των παιδιών και των νέων. Θα αφογκραστώ τις ανάγκες σας. Και τώρα θα πρέπει να ε, αναφέρω ότι ο δρόμος για την συνεννόηση και την αποδοχή ε, των δικαιωμάτων του παιδιού ήταν μακρύς και δύσκολος. Γιατί για αιώνες ολόκληρους είχε η άποψη ότι τα παιδιά ήταν ιδιοκτησία των ενηλίκων. Έγινε τιτάνια προσπάθεια και τεράστιο έργο ώστε να συνειδητοποιήσουν οι ενήλικες ότι και τα παιδιά είναι άνθρωποι και έχουν δικαιώματα. Πριν από 30 χρόνια ε, υιοθετήσαμε μια ιστορική απόφαση και ως ενήλικες υιοθετήσαμε τεράστιες ε, δεσμεύσεις για να εφαρμόσουμε τα δικαιώματα του παιδιού. Και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή τη σύμβαση που άλλαξε την πραγματικότητα για πολλά παιδιά. Η θέσπιση και η έγκριση της σύμβασης ήταν μια πραγματικά εξαιρετική εξαιρετική πολιτιστική, ένα εξαιρετικό πολιτιστικό επίτευγμα που έδωσε ελπίδα για σωστή αντιμετώπιση των ανήμπορων και ανυπεράσπιστων μέχρι στιγμής παιδιών και νιώθω ιδιαίτερα περήφανη γιατί είμαι Πολωνέζα. Ε, η χώρα μου ήταν πρωτεργάτη ε, τη προσπάθεια για την έγκριση αυτή τη σύμβαση. και είμαι περήφανη γιατί στη δική μου πατρίδα, την Πολωνία, το 1978 γεννήθηκε αυτή η ιδέα τη δημιουργία ενό ε, διεθνού οργάνου, μια διεθνού σύμβαση. Δεν θα είχαμε αυτή τη διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού αν δεν υπήρχε αυτό ο διαπρεπή Πολωνός Παιδαγωγό και γιατρό που ανέφερε η κυρία Κέμπα πριν από ο Γιάννους Κόρτσακ. Χάρη σε αυτόν και στις ε, καταπληκτικές παιδαγωγικές του απόψεις, Φτάσαμε σήμερα στις νομοθετικές διατάξεις της Σύμβασης. Ο Γιάννος Κόρτσακ ήταν αυτός που πρώτος έδωσε μάχη για να είναι το παιδί υποκείμενο δικαιωμάτων έλαβε ε, υπόψη τα παιδιά και τα δικαιώματα των παιδιών και υπενθύμησε στους ε, ενήλικες ότι θα πρέπει να δείχνουν σεβασμό προς τα παιδιά γιατί τα παιδιά δικαιούνται αυτό το σεβασμό. Και μέσα σε 30 χρόνια από τη στιγμή της υιοθέτηση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίναμε μάρτυρες πολλών θετικών αλλαγών. Και αναφίβολα ο κόσμος έγινε πιο ευνοϊκός για τα παιδιά. Εμείς όμως οι ενήλικες έχουμε λόγο για απόλυτη ικανοποίηση είναι τα πράγματα τόσο ιδανικά ώστε να μπορούμε να κοιμόμαστε ήρεμοι ότι τα παιδιά τη χάνουν προστασίας. Όχι, το αντίθετο. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού μας δείχνει την άγουσα που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Αλλά τα συμβαλόμενα μέρη θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Για να υλοποιηθούν όλες αυτές οι νομοθετικές διατάξεις θα πρέπει να αναλάβουν δράση οι ενήλικες και μόνο η κύρωση της συνθήκης δεν επιλύει τα προβλήματα των παιδιών ούτε καταργεί τις αδυναμίες της σχέσης μεταξύ του κόσμου των παιδιών και του κόσμου των ενηλίκων. Πολλά θα πρέπει να κάνουμε ακόμη για να δώσουμε σάρκα και οστά στη σύμβαση. Και με την τήρηση των διατάξεων αυτών και το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες και δεν μπορούμε να κοιμόμαστε ε, ήρεμοι και ανενόχλητοι στο μέτρο που η πείνα και οι ένοπλες σειράξεις σκοτώνουν πολλά παιδιά. Εκατομμύρια παιδιά ζουν σε απόλυτη εξαθλίωση, εξαναγκάζονται σε δύσκολες εργασίες, δεν έχουν πρόσβαση σε παιδεία και υγεία. Δεν μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι όταν χιλιάδες παιδιά είναι θύματα εγκληματιών. Οι στατιστικές μας δείχνουν ότι 25 εκατομμύρια παιδιά απειλούνται από φτώχεια αυτό είναι πραγματικά συγκλονιστικό, είναι πραγματικό σκάνδαλο. Θα πρέπει πάρα αυτά να εγγύψουμε στο πρόβλημα αυτό και να αντιστρέψουμε αυτές τις μακάβριες στατιστικές. Η 30η επέτειος της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι μεγάλη γιορτή, αλλά θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ο δρόμος μπροστά μας είναι μακρύς και δύσκολος. Θέλουμε κοινέ δράσεις για να αλλάξουμε την πραγματικότητα και να υλοποιήσουμε τους στόχους ε, τους στόχους που κατοχυρώνονται στη συνθήκη για τα δικαιώματα του παιδιού. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι εμείς οι ενήλικες είμαστε υπεύθυνοι να υλοποιήσουμε στο έπακρο τα δικαιώματα του παιδιού και να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ανάγκες του παιδιού. Και τώρα στρέφομαι στους συναδέλφους ε, ευρωβουλευτές. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερη στιγμή, στην αρχή της κοινοβουλευτικής θητείας, ε, στην αρχή της, της εντολής και της θητείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή, να βρούμε την πολιτική βούληση για να συνδέσουμε τα δικαιώματα του παιδιού με τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γιατί πολλές ε, σημαντικές διατάξεις είχαμε σε νομοθετικό επίπεδο. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε λοιπόν την πολιτική στιγμή ε, και την, ε, την ε, ειδική δυναμική αυτή τη στιγμή και να δημιουργήσουμε την πολιτική βούληση. Επίση, να συνεργαστούμε με τα άλλα θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με διεθνεί οργανώσει, με την κοινότητα των πολιτών και πρώτα απ' όλα να συνεργαστούμε με τα ίδια τα παιδιά και του νέου. Γιατί θα πρέπει να ακουστεί η φωνή των παιδιών. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές του πάνελ και κυρίως τους νέους που έλαβαν μέρος στη διάσκεψη αυτή. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την γλαφυρή παρουσίαση των εμπειριών σας και των απόψεών σας, γιατί δώσατε πραγματική αξία και αξιοπιστία στη συζήτηση με την παρουσία σας και τις μαρτυρίες σας. Και θα ήθελα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να σας ευχαριστήσω. Και να σας ευχαριστήσω και εκ μέρους του Αντιπροέδρου Φάμπιο Καστάλτο και σας προσκαλώ στην έκθεση Cartooning for Peace που θα γίνει που λαμβάνει χώρα στην στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε ντυθεί στα γαλάζια χρώματα ε, για να θυμηθούμε όλοι την ε, υιοθέτηση της σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που έγινε πριν 30 χρόνια και σε συνεργασία με τη UNICEF. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας. Εγώ σας ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε μια στιγμή γιατί πάντα μπορούμε να βελτιώνουμε τα πράγματα. Θα σας πρότεινα το εξής, γιατί παίρνω μηνύματα από τους νέους που λυπούνται που δεν μπόρεσαν να πάρουν το λόγο. Και σίγουρα έχετε δίκιο και δεν δώσαμε αρκετό χρόνο στους νέους για τη συζήτηση για να εκφραστούν. Σας προτείνω να κάνετε εσείς τις προτάσεις σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σε σχέση με τα όσα κάναμε σε αυτή την εκδήλωση να μας κριτικάρετε γιατί με την κριτική βελτιωνόμαστε ε, να μας κάνετε προτάσεις για του χρόνου του χρόνου θα τα ξαναπούμε θα ε, κάνουμε και έναν απολογισμό των όσων μας ζητήσατε και θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε και να σας δίνουμε περισσότερο το λόγο μην διστάσετε λοιπόν κάντε το και σας ευχαριστώ πολύ